Okay, good morning. Um, I think we, we, ought, we ought to make a start because I think... Νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε γιατί όσοι έπρεπε να έχουν έρθει έχουν ήδη έρθει. Παρόλο που καθυστερώντας μπορούμε να συζητάμε μεταξύ μας και αυτό είναι επίσης χρήσιμο. Τέλος πάντων, πρώτο θέμα στην ημεριστηριάτηση διάταξη για σήμερα είναι το νούμερο 6. Συνέχεια πρέπει να δοθεί στην εκχώρηση των νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών επί της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. Αυτή είναι μια έκθεση που είχε ξεκινήσει από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Ε, η οποία εξέτασε την ε, εφαρμογή των άρθρων 2.19 και 2.20 για τις ε, κατεξουσιοδιώτες και τις εκτελεστικές πράξεις ε, της, ε, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα διαδικαστικό θέμα. Θα σας ενημερώσω για τις συζητήσεις σχετικές που είχαμε στη διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Είναι διαφορετικό αυτό που είχε συμβεί από επιτροπή σε επιτροπή. σε κάθε περίπτωση ήταν διαφορετικό το κατά πόσο το κοινοβούλιο κατάφερε να αποσπάσει αυτό που ήθελε, δηλαδή σε ορισμένες περιπτώσεις που επιδίωξε να αντικατασταθούν οι, πράξεις, οι εκτελεστικές πράξεις με κατεξουσιοδότηση πράξη έτσι ώστε να έχει ε, λόγο το Κοινοβούλιο. Σε γενικές γραμμές η ε, Επιτροπή η δική μας ε, κατά οικονομικής και νομισματικής πολιτικής έχει καταφέρει αυτά που επεδίωκε και στην έκθεση που έχω συντάξει εξηγώ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσαμε και πώς αξιοποιήσαμε και την εμπειρία από τις εποπτικές αρχές. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι ότι χρειάζεται διαφάνεια από την πλευρά της Επιτροπής όσον αφορά την το, το χρονοδιάγραμμα για την υιοθέτηση των πραξιών κατά εξουσιοδότηση έτσι ώστε να μπορεί και το Κοινοβούλιο εγκαίρως να ασκεί το δικαίωμα ελέγχου του. Ορισμένε φορέ, για παράδειγμα, μπορεί μια τέτοια πράξη να εκδοθεί λίγο πριν τι διακοπέ και να μην έχουμε το χρόνο στη διάθεσή μα που θα έπρεπε για να τη συζητήσουμε. Υπάρχει επίση το ζήτημα των περίοδων των διακοπών. Ένα θέμα που συχνά θέτω στην διάσκεψη των Προέδρων είναι μεγάλο πρόβλημα για μας και ιδιαίτερα τώρα που θα έχουμε και τις ευρωεκλογέ το 2014 θα θέλαμε η Επιτροπή να μην εκδώσει πράξεις εκείνη την περίοδο γιατί η Επιτροπή η δικιά μας αλλά και γενικότερα δεν θα είναι διαθέσιμη να τις συζητήσεις Παρ' όλα αυτά, ε, μάλλον θα είναι αναγκαστικό κάποια πράγματα να εκδοθούν, κάποιες πράξεις να εκδοθούν. Φαντάζομαι κάτι αντίστοιχο θα συμβαίνει και όσον αφορά την Ολομέλεια. Τουλάχιστον θα πρέπει να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία, να μην ε, εκδοθούν πολλές πράξεις εκείνη την περίοδο. Υπάρχουν κάποιες τροπολογίες από τους σοσιαλιστές, εννέα τον αριθμό, και ο κύριος Αντολίν έχει υποβάλει τροπολογίες σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλες τροπολογίες. Σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είναι αποδεκτές. Ε, πριν να δώσω το λόγο σε εκείνους που έχουν προτείνει τροπολογίες, Θα ήθελα να ρωτήσω κάποια πράγματα για συγκεκριμένες διατυπώσεις. Ε, στην τροπολογία 3, για την παραγραφο 2, καταλαβαίνω τι προσπαθείτε να πείτε. Αυτό που προσπαθούσα εγώ να καλύψω είναι ότι είχαμε κάποιες πληροφορίες από την ΕΣΜΑ. Ότι τη μέσω των ιδεολογικών σκέψεων δύναμη τις απαιτούμενες πληροφορίες και την απαιτούμενη καθοδήγηση. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε τώρα, να πάρουμε τη δική σας διατύπωση ίσως και να προσθέσουμε κάποια ακόμα στοιχεία για να είναι ότι θα υπάρχει η απαιτούμενη κατεύθυνση για τις σημαντικές επιλογές πολιτικής. τροπολογία 7, κύριος Μάρτιν, ζητά να αποστέλλεται γραπτό σε όλα τα μέλη της Επιτροπής τα στοιχεία αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι υπερβολικό. Καταλαβαίνω τι επιδιώκεται, ότι θα πρέπει όλοι να είναι ενήμεροι, Και όντω θα ήταν βέλτιστη πρακτική και θα ήταν καλύτερο η γραμματεία να κυκλοφορεί αυτά τα στοιχεία σε όλα τα μέλη. Υπάρχει μια άλλη πρόταση, τουλάχιστον να κυκλοφορούνται αυτά τα στοιχεία στον εισηγητή και στους ε, σκιώδεις. θα μπορούσαμε λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό. Ο κύριος Μάρτιν δεν είναι εδώ, αλλά θα σχολιάσω την τροπολογία του, την 9. Ε, θεωρεί ότι η προθεσμία των δύο μηνών για την ε, διοργανική συμφωνία, ε, συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι υπερβολικά μικρή και προτείνει να το διαγράψουμε. Θα μπορούσε να γίνει αυτό αλλά θα ήθελα να επισημάνουμε ότι αυτή η προθεσμία των δύο μηνών μπορεί να είναι πολύ μικρή, ιδιαίτερα όταν το ζήτημα είναι περίπλοκο ή εκτεταμένο. Αν το για την διατύπωση της τροπολογίας 13, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Είναι μάλλον γλωσσικό το θέμα στα αγγλικά. θα πρέπει να καταστήσουμε σαφές τέλο πάντων είναι ότι εκείνη την περίοδο θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία που να λειτουργεί. Στην 15 προτείνεται τη λέξη address και αναρωτιέμαι αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρευρίσκονται, να, γίνεται μια ακρόαση και να παρευρίσκονται στην Επιτροπή για να εξηγούν τη θέση τους. Πιστεύω ότι αυτό που θα έπρεπε να είναι, να είναι ένα διαθέσιμη, να βρίσκεται στη διάθεσή μας, και να μας ενημερώνουν αν χρειαστεί. Επομένως, ίσως κάπως να αλλάξουμε τη διατύπωση για να γίνει αυτό πιο σαφές. Και τέλος, ανέφερα το ζήτημα stakeholder appointment του ορισμού των ενδιαφερόμενων στο κείμενό μου, γιατί το θεωρώ σημαντικό, ακόμα και αν δεν έχει άμεση σχέση με τις κατεξουδότητες συμπράξεις, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να το αναφέρουμε. Πρέπει αυτός ο ορισμός, ο καθορισμός να γίνεται μέσα σε ένα σωστό χρονοδιάγραμμα, γιατί διαφορετικά απλώς ε, καταλήγουμε στους συνηθείς υπόπτους να συμμετέχουν κάθε φορά. Αυτά είναι τα σχόλια που είχα να κάνω σε σχέση με τις τροπολογίες που υποβάλατε και σας ευχαριστώ για αυτές. Εάν οποιοδήποτε θα ήθελε το λόγο τώρα για να διευκρινίσει οτιδήποτε. Thank you very much, uh, Sharon, for... Ευχαριστώ πολύ, Σάρον, για την εισαγωγή σου. Θα εξηγήσω πάρα πολύ σύντομα τις τροπολογίες που δεν είναι ακριβώς τροπολογίες, μάλλον προτάσεις μου είναι. Γιατί η πρόθεσή μου είναι να καταλήξουμε σε ένα συνετικό κείμενο, να το κοιτάξουμε, να συμφωνήσουμε, ορισμένα είναι γλωσσικά τα στοιχεία αυτά και είμαι πεπισμένος ότι η συγγήτρια κατέχει πολύ καλύτερα την Αγγλική από τον υποφαινόμενο. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω το εξής πρώτο τα ε, regulatory technical standards που έχουμε τα αριθμιστικά πρότυπα είναι μια ειδική κατηγορία κατεξοδότηση πράξη. Και είναι κατεξοδότηση πράξη ή μπορεί ε, να υπάρξουν και κάποιες ξεχωριστές κατεξοδότηση πράξης. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρξει μια παρεξήγηση, δηλαδή να μην θεωρήσουμε ότι τα πρότυπα αυτά δεν είναι κατεξοδότηση πράξης. Είναι τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και θα πρέπει οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να επιληφθούν του θέματος και μάλιστα είναι πάρα πολύ ειδική αυτή και συγκεκριμένη διαδικασία. Λοιπόν, καταρχήν θα μπορούσαμε να έχουμε άλλες κατεξοδότηση πράξεις τεχνικής φύσεως ας πούμε που θα πρέπει να υπάρχει και εκεί ε, αξιολόγηση. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεύτερον, τα σημαντικά στοιχεία. Η ουσιώδη ή μη ουσιώδη στοιχεία. Το θέμα είναι να δούμε τι μέσο είναι αυτό. Είναι νομοθετικό, είναι ε, εξουσιοδότηση, πράξη ή εκτελεστική. Και έχω μια τροπολογία που ε, είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί ε, σύμφωνα με τη συνθήκη είναι θέμα του νομοθέτη. Ο νομοθέτης δεν μπορεί να εκχωρήσει αυτή την αρμοδιότητα σε κανέναν ούτε να, εξουσιοδοτήσει κανένα άλλο μηχανισμό ή καμιά άλλη αρχή. Αυτό σημαίνει. Στη Frontex υπάρχει ολόκληρη απόφαση του δικαστηρίου ε, που προσεγγίζει τα ουσιώδη στοιχεία και τα σημαντικά και λέει ότι ουσιώδη στοιχεία είναι αυτά που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη και εξέλιξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή αυτά που ορίζουν τους μεγάλους πολιτικούς στόχους και τις μεγάλες κατηγορίες δαπανών, τις μεγάλες πολιτικές κτλ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια ουσιώδη στοιχεία που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του νομοθέτη. Αυτά δεν εκχωρούνται, δεν ε, ε, διαβιβάζονται, δεν μεταβιβάζονται κτλ. Υπάρχει κάτι άλλο όμως που μπορεί να εκχωρηθεί στα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα, ε, αλλά σε αυτό το στοιχείο εγώ θα ήθελα να τονίσω ε, την ευθύνη του ε, νομοθέτη να έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για τη ρύθμιση των ουσιοδών στοιχείων. Είναι δουλειά της νομοθετικής εξουσίας αυτή και ευθύνη μας στη δημοκρατία. Και νομίζω το άρθρο 90 είναι σαφές και θα πρέπει να το τηρήσουμε κατά γράμμα. Τα ουσιώδη στοιχεία δηλαδή ε, ποια είναι αυτά και ε, η κατεξοδότηση πράξης ε, είναι συμπληρωματικές, παραπληρωματικές ή δεν αφορούν ουσιαστικά στοιχεία παρά μόνο δευτερεύοντα. Να τα ξέρουμε αυτά, να τα ξεκαθαρίσουμε στο μυαλό μας. Επίσης, για τους μηχανισμούς ευελιξίας προτείνω ένα κριτήριο που μου φαίνεται χρήσιμο το έχω προτείνει και σε άλλη επιτροπή που ήμουν εισηγητής για αυτό το θέμα. Ε, σε όλες τις επιτροπές αυτές θα πρέπει να υπάρχει κάποιος αρμόδιος για να υπάρχει μια στοιχειώδη και καλύτερη δυνατή συνοχή ανάμεσα στις διάφορες επιτροπές. Δεν ξέρω ποιος αν αυτός, κάποιο μέλος του Προεδρείου ή Πρόεδρος κτλ. Ε, για να υπάρχει μια ενιαία και κάπως συνεκτική αντιμετώπιση και συνεπής από επιτροπή σε επιτροπή. Και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον ο κάθε ε, εισηγητής ε, νομοθετικής έκθεσης να παρακολουθεί την εξέλιξη. Γιατί ο εισηγητής είναι κατεξοχήν ο πλέον αρμόδιος για αυτά τα θέματα, έχει μελετήσει το κάθε θέμα σε μεγαλύτερο βάθος και νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο. Τα υπόλοιπα είναι γλωσσικά τα υποβάλλω στην εισηγήτρια για να τα κοιτάξει και όσο γίνεται περισσότερο να φροντίσει να μπουν στην έκθεση. Προφανώς δεν θα τις καταθέσω, δεν θα τις καταθέσω τις τροπολογίες μου μονομερός. Ε, παρακαλώ την εισηγήτρια να τις συμπεριλάβει όσο γίνεται σε συμβαστικές προτάσεις και να καταλήξουμε σε συνενετική έγκριση του κειμένου, να συμφωνούν όλα τα μέλη. Ευχαριστώ, Αντολίν. Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρουμε. Βέρνερ, συγγνώμη, είχα ανοίξει λάθος κατάλογο και δεν είχα δει ότι είσαι για το ΕΛΚ. Ε, εγώ να δεις. Σήμερα το πρωί το έμαθα ότι είμαι σκιώδης συγγετής για το ΕΛΚ. Ε, δεν το ήξερα, το ανακαλύπτω κι εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Σάρων πραγματικά έχει συμπεριλάβει τα σημαντικότερα στοιχεία στο σχέδιο έκθεσή της. Θυμάστε το ΕΜΙΡ, στην αρχή του έτους τα ίδια είχαμε ζήσει. Πάρα πολύ μικρές ε, ήταν οι προθεσμίες, πολύ γρήγορα έφεραν κατ' εξουδότηση πράξης και δεν μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο. Τι μας είπε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κυρία Χέντεγκάρτ, εξ ονόματος όλης της Επιτροπής, δήλωσε ότι στο μέλλον Πρώτον, θα είναι κοντά μας χρονικά και ε, θα μας ενημερώνει και θα έχουμε αρκετό χρόνο για διαβουλεύσεις και στην ίδια τη διαδικασία θα μας συμπεριλαμβάνει καλύτερα. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος, πλην όμως το ερώτημα είναι αν καταφέρουμε όχι μόνο στην Επιτροπή μας αλλά σε όλο το Κοινοβούλιο το θέμα των κατεξουδότησης νομικών πράξεων ε, να μπορούμε να το αξιολογούμε σωστά. Και θέλω πραγματικά να πω ότι έχει δίκιο η Σάρον στις παρατηρήσεις της πρώτον το κοινοβούλιο που είναι συνομοθέτης θα πρέπει να φροντίσει όσο γίνεται τα σημαντικά, τα ουσιώδη στοιχεία να είναι ε, στο ουσιαστικό κείμενο, στο νομοθετικό κείμενο και όχι στο δευτερογενές. Ε, δεύτερο. Το είπε και η Σάρων προηγουμένως, η διαφάνεια θα πρέπει να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη. Δηλαδή να γνωρίζουμε χρονικά όλα αυτά πώς προγραμματίζονται, γιατί έχουμε το δικαίωμα να έχουμε ακριβώς με διαφάνεια ένα χρονοδιάγραμμα που μπορεί καμιά φορά να καθυστερεί και να παρατείνεται. Αυτά τα γνωρίζουν οι πάντες, συμβαίνουν. Αλλά γενικά η πρόταση της Προέδρου μπορεί να είναι η βάση για μια καλή γνωμοδότηση. Και αυτό που πρότεινε ο συνάδελφος Σάντσες Περσέδο το γνωρίζουμε. Θα πρέπει να τα πούμε ο καθένας στην ομάδα του. Μέχρι τώρα δεν το έχουμε κάνει. Και εκεί που έχει νόημα ε, υποστηρίζουμε βέβαια και όσα λένε οι σοσιαλδημοκράτες, αλλά ευθυγραμμιζόμαστε 100% ε, πίσω από την εισηγήτρια, την κυρία Σάρον Μπόλς. Ευχαριστώ, Βέρνερ. Τα περισσότερα από αυτά που μας είπε ο Άντολιν τελικά θα τα καταφέρουμε νομίζω σύν το χρόνο. Έχουμε και διάφορες διμερείς συμφωνίες ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το επίπεδο που δεν έχει συνολικά το Κοινοβούλιο και ξέρετε οι προηγούμενες συμφωνίες δεν θα πρέπει να υπεσκελιστούν από μια γενική συμφωνία Αυτό θα μας προκύψει από το πουθενά από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Σβέν. Ουσιαστικά το μόνο που έχω να πω είναι ότι καλωσορίζουμε την έκθεση σου Σάρων. Οι τροπολογίες των συναδέλφων μπορούν να γίνουν αποδεκτές ε, από την ομάδα μας. Υπάρχει ένα θέμα που ανέφερε και εσύ στι εισαγωγικέ σου παρατηρήσει. Ε, πρόκειται για την τροπολογία Μάρτιν. Κατανοούμε την ανησυχία που εκφράζει. Ταυτόχρονα η τροπολογία 5 της ΚΕΙ καλύπτει με πιο ικανοποιητικό τρόπο το θέμα, επιτυγχάνει τον ίδιο σκόπο, σκοπό που θέτει και ο Μάρτιν ε, και δικαίως θέλει επιθυμεί όλα τα ανεξάρτητα μέρη να ενημερώνονται για τη διαδικασία, αλλά μπορούμε να το κατοχυρώσουμε με τον τρόπο που προτείνει και η τροπολογία 5. Πάντως, ε, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση Και δεν συντρέχει λόγος, ε, Σάρων, ε, για να μην συμπαραταχθούμε κι εμείς. Okay. Ευχαριστώ. Και εγώ λιγοστά έχω να προσθέσω. Είναι κέρια σημασίας να ορίσουμε τη διαδικασία βάση των οποίων θα λειτουργήσουν τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και πράξη κατά εξουσιοδότηση και οι σχέσει ανάμεσα στι συναρμόδιε επιτροπέ, αλλά και τι εθνικέ αρμόδιες αρχέ. Είναι ίσονο σημασία στις τροπολογία μου. Φέρνουν επί τριών ζητημάτων. Πρώτον, ανταλλαγή πληροφοριών και ενημέρωση, μόλι το ανέφερε ο Σβέν. Και ελπίζω με την τροπολογία 5 να καλύπτω όλε τι πολιτικέ ομάδε για να επιτύχουμε ε, διευρυμένη διανομή από τη γραμματεία όλων των εγγράφων. Άλλο βασικό ζήτημα είναι η συνοχή, η συνέχεια μετά τις εκλογές και μετά την πρώτη φάση αυτού του άπειρου αριθμού των κατεξουσιοδότηση πράξεων. Αυτή η διαδικασία πρέπει να συνεχιστεί μετά τις εκλογές διότι μπορεί να μην επανέλθουμε σε κάποια ζητήματα οπότε μετά τα αποτελέσματα τη εκλογική αναμέτρηση πρέπει να μάθουμε ποιο θα είναι αρμόδιο για κάθε επιμέρου θέμα και να μεριμνήσουμε ώστε να διορίσουμε ένα νέο εισηγητή για τι πράξει κατά εξουσιοδότηση, αν πολιτική ομάδα. Οπότε, εάν επιτρέψουν κάποιοι σκιώδει, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κάθε πολιτική ομάδα επισήμω θα διορίσει κάποιον και δεν θα μείνει κενή η θέση. Και αν, κάποιος ε, δεν, είναι, αν δεν υπάρχει κάποιο αρμόδιο για κάθε θέμα, θα χάσουμε ε, την μπάλα. Δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε την διαδικασία διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να επισημοποιηθούν, να θεσμοθετηθούν τέτοιου είδους διαδικασίες και ε, μετά τη σύσκεψη με την ομάδα ΕΣΜΑ ε, ήμουν πολύ ικανοποιημένη. Ήρθαν πριν από λίγες εβδομάδες για να μας μιλήσουν για την ε, περχόμενη φάση διαβουλεύσεων και ελπίζουμε να συνεχιστούν. Έχουμε αποστείλει και εμείς σχόλια. Ελπίζουμε να έχουμε την επιθυμητή έκβαση σε σχέση με τα προσδοκόμενα και το βασικό είναι να επισημοποιηθεί αυτό για να μπορέσει να προχωρήσει η διαδικασία ε, και να εξασφαλιστεί λοιπόν η συνέχεια με τη νέα θητεία, με το νέο κοινοβούλιο ε, στο σωστό επίπεδο και εν ευθέτω χρόνο ε, να εξασφαλίσουμε τη συνοχή και τη συνέχεια της διαδικασίας. Ε, με αυτά τα σχόλια δεν έχω τίποτα να προσθέσω επ' αυτού. Τροπολογία 15 τώρα. Βλέπουμε ότι όταν το ζητάει η αρμόδια επιτροπή θα πρέπει να ε, ε, προσέρχονται ε, το να προβλεφθεί θεσμικά η δυνατότητα να έρχονται ενώπιον της Επιτροπής ε, πιστεύω ότι είναι για να καταλήξουμε τελικά σε συμβασμό μέσω της τροπολογίας 15. Ευχαριστούμε Πρόεδρος και ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Όχι, ωραία, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και νομίζω πως η ΚΕΙ είπε αυτά που σκεφτόμουν, πως πρέπει να κινηθούμε σε σχέση με την τροπολογία 15. Όταν θέλουμε θα πρέπει να μπορούν να έρχονται, δηλαδή θα τους καταναγκάσουμε κιόλας. Γνωρίζετε ότι ορισμένες φορές υπάρχει, υπάρχουν χρονικά προβλήματα για αυτή την ενημέρωση. Μπορώ να πω στους συντονιστές ε, τι πρέπει να κάνουν. Αλλά σε μια πρώτη συνεδρίαση που κάναμε στην τωρινή θητεία με τους συντονιστές είχαμε πει ότι θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με τα μέτρα δευτέρου επίπεδου για τη φερεγγιότητα 2 και τα λοιπά και ο Πίτερ Σκίνερ ήταν ακόμη εδώ και επέμεινε και εκείνο ότι πρέπει να συνεχίσει η ίδια ομάδα να επιλαμβάνει του ζητήματος. Η ομάδα των εισηγητών, αν μπορώ ε, να την αποκαλέσω έτσι, δεν υπάρχει ως τέτοια πλέον και ω εκ τούτου πρέπει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για να πάρουμε απόφαση. Μπορούμε να το αναφέρουμε, αλλά δεν, ε, ε, ακόμη και αν δεν το κρίνει ενδεδειγμένο η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Εφόσον όμως μιλάμε για διοργανικά ζητήματα και όχι για αρμοδιότητες εμμονωμένης επιτροπής, με κάποιο τρόπο θα μπορέσουμε να βάλουμε και αυτό το σχόλιο θα κυκλοφορήσουν ε, σχέδια συμβαστικών τροπολογιών, αλλά πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ε, τροπολογιών ε, θα εγκριθούν τελικά ή θα συγχωνευτούν όταν υπάρχει επικάλυψη. Ευχαριστούμε. Κλείνει αυτό το σημείο. Έχω μεταθέσει το σημείο 7. Την έκθεσή μου δηλαδή για την αποκάλυψη πληροφοριών μη οικονομικής φύσεως. Υπάρχει ένα διαθέσιμο προσχέδιο, όπως είπα σε μερικούς. Το πρόβλημα είναι πώς, ποιος είναι ο σωστός μορφότυπος ε, έχει αναβάλει τη συζήτηση και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και θα το εκμεταλλευτούμε κι εμείς για να μπορέσουμε να εργαστούμε ε, παραπάνω προτού ε, δημοσιοποιήσουμε τη δική μας γνωμοδότηση. Και έτσι φτάνω στην επανεξέταση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Ο εισηγητής μας είναι ο Σβέν Γκίγκολτ. Σβέν. Μήπως να ξεκαθαρίσουμε ε, ότι ε, αρχίσαμε νωρίς το θέμα και μας λείπουν σκιώδεις ηγητές. Τώρα δεν ξέρω αν ο Ροφ Κλίντς είναι εδώ στο κοινοβούλιο, ο Βολφ Κλίντς. Είναι κρίμα. Κάτι απαντάει ο βοηθός του. Να περιμένουμε πέντε λεπτά να έρθει ο Βολφ Κλίντς. Δεν ξέρω κυρία Πρόεδρε, εσείς τι φρονείτε σχετικά. Νωρίς το ξεκινήσαμε. Θα πρέπει να το συζητήσουμε παρόντων των σκιωδών. Uh, δεν πειράζει. Να καθυστερήσουμε λίγο. 9 και 25 όμως λέει ενδεκτικά ότι θα αρχίζαμε. Ναι, αλλά η βοηθή του Βολφ μας λένε ότι σε 5 λεπτά έρχεται. Σε μια μυστική γλώσσα μου το είπε, δεν το άκουσες. Α, κατάλαβα, του στείλε SMS. Όχι, όχι, γερμανικά εννοώ, Βρεσάρων. Uh, so wait. I, I, I agree with you that it's better. Ναι, ναι, συμφωνώ. Πέντε λεπτά διάλειμμα. Νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε, Σφεν, έτσι σιγά-σιγά. Θα τα σημειώσουν οι βοηθοί του Βόλφ Klintz αυτά ή μέχρι να έρθει. Καλά. Äh, λοιπόν, εισαγωγικά για τη συζήτηση αυτή θέλω να πω το εξή εξ αρχή Η συζήτηση αυτή για τη χρηματοπιστωτική εποπτεία μας συνοδεύει από την αρχή της θητείας. Από την αρχή, αρχή είχαμε πολύ μεγάλες πλειοψηφίες ε, για το θέμα αυτό, για να το συζητήσουμε. Το πρόβλημά μας δεν ήταν ότι είχαμε μεγάλες διαφορές μεταξύ μας στο Κοινοβούλιο τουλάχιστον όχι σε μεγάλο βαθμό. Αλλά κάναμε μεγάλους καυγάδες με το Συμβούλιο. Σε ποιο βαθμό χρειαζόμαστε και σε ποιο βαθμό θα έχει δικαιώματα μια ενιαία χρηματοπιστωτική εποπτεία. Θυμάστε, τότε είχαμε μια έκθεση του Jacques Delors την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μεγάλο βαθμό υιοθέτησε και κατέθεσε δική της πρόταση. Ακολούθησε μακρά διελκυνσίδα με το Συμβούλιο και μετά το Συμβούλιο ε, δεν ήθελε να ξέρει τίποτα μετά την κρίση για πολλά από τα όσα είχε αποφασίσει από την έκθεση Ντελαροζιέ. Ορισμένα επεδείχθηκαν χρήσιμα και υλοποιήσιμα και κάποια άλλα ζητήματα ε, θέτουν ερωτηματικά. Καλό είναι λοιπόν να τα συζητήσουμε, να δώσουμε και ένα input, τη δική μας πρόταση στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχει βέβαια αλλάξει το τοπίο έκτοτε, διότι απλούστατα έχουμε κοινή εποπτεία των τραπεζών και στην Ευρωζώνη και για τις υπόλοιπες χώρες και αυτό πραγματικά δημιουργεί κάποια ερωτηματικά για τα υπόλοιπα και για την υπόλοιπη χρηματοπιστωτική εποπτεία. Ορισμένα θα φανούν στην πορεία, αρκεί να σκεφτούμε ότι μόλις εχθές μάθαμε πόσο έχουν προχωρήσει ε, οι εργασίες στο SSM, ε, στον ενιαίο μηχανισμό εποπτείας ε, παρόλο που αποφασίσαμε πρόσφατα ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για το εγχειρίδιο θα έχει ε, τον πρώτο λόγο, αυτή η ένταση και ο διαπλεκτισμός θα μεταφερθεί και σε άλλους τομείς και θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Σε όλο και περισσότερους τομείς και σε όλο και περισσότερες χώρες ε, παγκοσμίω ε, γίνεται μια προσπάθεια προς ένα διτό σύστημα. Δηλαδή και τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες ε, είναι στην ίδια εποπτεία στο ίδιο σημείο και από την άλλη μια εποπτική αρχή που εποπτεύει τις χρηματαγορές για την προστασία των επενδυτών και για αποτελεσματικές χρηματαγορές. Αυτά τα θέματα Λοιπόν, το λεγόμενο Twin Peak μέχρι τώρα δεν το έχουμε συναντήσει εδώ και ε, στο θέμα της ε, τραπεζικής εποπτείας στον νέο εποπτικό μηχανισμό έχουμε το ζήτημα ε, των ασφαλιστικών εταιριών που λόγω της νομικής βάσης εξαιρούνται τελείως. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει. Ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Είναι όλη η συζήτηση μερώνει. Δηλαδή, θα πρέπει να κοιτάξουμε τι γίνεται με το σορτάρισμα, με τις ακάλυπτες ε, πωλήσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα λέει το δικαστήριο, γιατί στη ε, νομοθεσία ο έχει περιορίσει τις εξουσίες. Εμείς δεν είμαστε οπαδοί αυτής της σκιασμερών μερών στο Κοινοβούλιο στο παρελθόν. Ούτε επί της ουσίας συμφωνούσαμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά τώρα, αν υπάρξει διευκρίνηση από το δικαστήριο που είναι πιο φιλική, να το πω, προς τη δημοκρατία και πιο ε, βολική, θα μπορούσαμε και εμείς να κάνουμε κάτι και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης δεν θα πρέπει να αρνείται να προχωρήσει. Το επόμενο ερώτημα που τίθεται κατά την άποψή μου είναι τι θα γίνει με την αξιολόγηση των ίδιων των εποπτικών αρχών. Πού θα πρέπει να εστιάσουμε σήμερα, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα μιας θεώρησης ε, και οι τρεις ΙΖΑ έχουν κάνει καλή δουλειά ε, σε πολλούς τομείς, έχουν γίνει μεγάλες πρόοδοι. Βλέπε ψηφοφορίες λέει, ψηφίζουν παρακαλώ και στις τρεις ε, και στον ESRB δεν είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής αλλά ψηφίζουν πραγματικά, γίνονται δημοκρατικές διαδικασίες εκεί και οι τρεις λοιπόν αυτές εποπτικές αρχές έχουν ε, τολμήσει πράγματα που δεν άρεσαν σε σημαντικούς φορείς της αγοράς. Αυτό είναι πρόοδος για την εσωτερική αγορά. Σκεφτείτε και μόνο την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ε, τι κάνει για τα τεστ κοπόσεως και τη βελτίωση ε, των ιδίων κεφαλαίων που έχουν πετύχει. Και το επόμενο θέμα βέβαια είναι λίγο σχετικό. Αν δούμε τα διάφορα καθήκοντα που έχουμε εμείς ως νομοθέτες ε, ε, αναθέσει στις τρεις αρχές για τη μικροπροληπτική εποπτεία πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτές οι αρμοδιότητες και αυτά τα καθήκοντα και εξουσίες που τους έχουμε χωρίσει δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ. Δηλαδή θα πρέπει να διαμορφώσουμε εμείς άποψη. Τι έγινε, δεν υπήρχε κρίση. Έχουμε δικαιώματα επέμβαση στη κρίση για τις εποπτικές αρχές. Τους έχουμε δώσει, δεν τα χρησιμοποίησαν καθόλου το περίφημο άρθρο 18. Επίσης έχουμε και το θέμα γύρω από την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ισχύει αυτό παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 28 κράτη στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ισχύει και εφαρμόζεται το κοινοτικό δίκαιο και τηρείται. Έχω κάποιες αφιβολίες εγώ. Ε, στα κράτη-μέλη ε, ε, κανονικά θα πρέπει να εφαρμόζεται και θα πρέπει να ανακαλούνται στα στην τάξη τα κράτη που δεν τις εφαρμόζουν. Το ίδιο ισχύει και για την υποχρεωτική ε, διευθέτηση και διακανονισμό διαφορών. Τι έγινε, συμφωνούν πάντα οι εποπτικές αρχές σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν αντιδρούν. Δεν μου φαίνεται πάρα πολύ αξιόπιστο. Και πραγματικά εκεί που αποδίδουν, παρόλο που έχουν μικρές καθυστερήσεις, είναι στις κατεξουδιώτηση πράξεις και την νομοθεσία. Αυτό πάνω κάτω λειτουργεί. Μπορεί να υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις είπαμε, αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους αυτές οι υπηρεσίες και θα πρέπει να ρυθμίσεις. Αλλά ακόμα και αυτό και αυτές οι αρμοδιότητες που τους εκχωρήσαμε ε, δεν ε, υλοποιούνται, δεν ασκούνται με το σωστό τρόπο ε, και γι' αυτό θα πρέπει να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Ένα από τα πιθανά συμπεράσματα είναι να πούμε η υπερβολική η διακυβερνητική συνεργασία, ε, πολύ μεγάλη ε, δυνατότητα άσκησης βέτο και τίθεται και ζήτημα πειθαρχίας απέναντι στις κυβερνήσεις και δεν έρχονται καν προσυζήτηση διάφορα θέματα αυτά στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Και τα δικαιώματα δηλαδή ε, επέμβασης που έχουν, οι κυβερνήσεις πολλές φορές δεν τα θέλουν. Έχω πάει στις διάφορες εθνικές εποπτικές αρχές και έχω συζητήσει εκεί με εργαζομένους και η πρόσβαση σε δεδομένα και σε στοιχεία δεν είναι δεδομένη παντού ε, αυτή, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Τους έχουμε δώσει μεγάλες ε, ε, αρμοδιότητες και εξουσίες μπορούν να ζητούν στοιχεία, ε, όλα να τα έχουν στη διάθεσή τους και τα κράτη πρέπει να τους τα δίνουν, είναι υποχρεωμένα. Βέβαια, αυτά τα δικαιώματα δεν τα χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου, διότι θεωρούν ότι στο Εποπτικό Συμβούλιο δεν το θέλουν αυτό οι ανώτεροι τους να γίνονται τέτοια ερωτήματα. Ε, και έτσι λοιπόν και η γάτα την ουρά της. Τους έχουμε δώσει λοιπόν δικαιώματα τα οποία ήδη δεν τολμούν να ασκήσουν ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και δεν έχουν και πλειοψηφία προς την κατεύθυνση αυτήν. Εξού και ε, σε αδράνεια οδηγούμαστε σε πολύ σημαντικές περιπτώσεις και τελικά λοιπόν έχουμε ένα κατακαιρματισμό της εσωτερικής αγοράς και ένα μεγάλο κίνδυνο, πώς να το πω, εμφανίζονται σημαντικές ε, τάσεις επανεθνικοποίησης και στην εποπτεία των χρηματαγορών. Και αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει σε βάση στο Κοινοβούλιο. Το ίδιο ισχύει και ε, με τη στελέχωση και τους πόρους που έχουν αυτές οι υπηρεσίες. Ε, ζητήσαμε ξεχωριστή πίστοση γραμμή στον προπολογισμό. Ο Βέρνερ Λάγκεν το ζήτησε στην περασμένη του έκθεση για τον προπολογισμό και εμεί επανειλημμένα το έχουμε ζητήσει και θα πρέπει να εμείνουμε όπως και στο παρελθόν. Και ένα τελευταίο. Οι μικροπροληπτικές εποπτικές αρχές είναι η μείωψη του νομίσματος. Έχουμε και τις μακρο προληπτικές εποπτικές αρχές. Τα ίδια ε, μπορούμε να διαπιστώσουμε εκεί. Η ESRB δεν είναι και το αγαπημένο παιδί, παρόλο που είναι πάρα πολύ αποφασιστική η μακροπροληπτική εποπτεία. Και σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση των χρηματαγορών, των χρηματοπιστωτικών, έχουν γίνει πολύ λιγότερες πρόοδοι εκεί. Υπάρχει η τάση πολλές φορές να ρυθμίζουμε τα πάντα μέχρι τελευταίας κεραίας για τα μικρά ζητήματα, αλλά για τα μεγάλα. Ε, τι γίνεται με ε, τις αντικυκλικές ε, ε buffer zone, τα μαξιλαράκια που μπορούμε να φτιάξουμε, την ενιαία λογιστική. Όλα αυτά δεν τα λέμε, αλλά λέμε τα πάρα πολύ μικρά. Η ESRB όμως στην νομοθεσία έχει κάνει σημαντικές νομοδοτήσεις που ε, αφορούν και συμπληρώνουν ε, με ενδιαφέροντα τρόπο την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Φεραγγιότητα 2 ας πούμε. Το επανέλαβε ο κύριος Δράγκη. Ε, είπαν ότι χρειαζόμαστε τελείως συμμετρικούς κανόνες για την απορρόφηση της πτυτικότητας των χρηματαγορών ή στις πιστώσεις σε ξένο νόμισμα να έχουμε πιο αυστηρές ρυθμίσεις και στην οδηγία για τις κεφαλαϊκές απαιτήσεις ε, και στη ΣΥΡΑ έχουν βάλει προϋποθέσεις και όρους αλλά οι προτάσεις τους δεν ήταν πάντα οι επιθυμητές. Ήταν οι πρώτοι που εκλήθησαν να ε, συμμετέχουν πλήρως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, πρέπει να κάνουμε και την αυτοκριτική μας εδώ. Στη νομοθετική διαδικασία δεν ελήφθησαν ε, σοβαρά υπόψη. Πώς μπορούμε λοιπόν να δούμε τη μακροπροληπτική εποπτεία που είναι συχνά πιο σημαντική από τη μικροπροληπτική, πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε στη νομοθετική διαδικασία και ε, να έχουν λόγο ουσιαστικό κατά τη διάρκεια της ε, διαδικασίας αυτής. Αυτά ε, είναι οι βασικότερες σκέψεις επί της ουσίας. Με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένω να ακούσω τις δικές σας απόψεις και θέλω την έκθεση αυτή πραγματικά να την κάνουμε σε ένα πνεύμα συνεργασίας στο Κοινοβούλιο. Να είναι ένα κοινό μας εγχείρημα γιατί είναι και βάση για την αναθεώρηση όπου θα έχουμε απέναντί μας το Συμβούλιο. Καλό είναι να έχουμε μία φωνή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Στους σκιώδεις τώρα θα πάω. Άστριτ, θέλετε λόγο. Μένα δεν θα με περίμενες. Oui, Madame la Présidente. Euh, moi, je remercie le rapporteur, M. Gugolt, Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για αυτές τις, αυτή την έκθεση. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι ίσως είναι νωρίς να λάβουμε θέση σε όλα αυτά τα ερωτήματα που τίθενται. Επομένως, εγώ δεν μπορώ να πάρω ε, θέση τόσο γρήγορα και επίσης γιατί ακόμα ε, αλλάζει αυτή η έκθεση και για πρακτικούς λόγους και για λόγους διαδικαστικούς. Πρόκειται η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας για τις Ευρωπαϊκές Ρυθμιστικές Αρχές που αυτή τη στιγμή μεταβάλλεται άρδιν. Και ε, το διαπιστώνουμε αυτό καθημερινά. Όταν δημιουργήθηκαν το 2010 αυτές οι ρυθμιστικές αρχές, υπήρχε μια ρήτρα η οποία έδινε την δυνατότητα, μάλλον ε, έδινε την υποχρέωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναφέρει το αργότερο μέχρι τον Ιανουάριο του 2014 ε, να προβάλλει μια έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας αυτών των αρχών. Και φαίνεται ότι η Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων αποφάσισε να προλάβει αυτήν την έκθεση της Επιτροπής και να καταρτήσει μια έκθεση δικής της πρωτοβουλίας. Δεν είμαι και λοιπόν ιδιαίτερα πεπισμένη ότι αυτό θα λειτουργήσει. Έχει γίνει Γίνεται μάλιστα ακόμα πιο ενδιαφέρον το θέμα όταν λάβουμε υπόψη μας ότι το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από μια εταιρεία συμβούλων να καταρτήσει ακόμα μια έκθεση για τον τρόπο λειτουργία αυτών των αρχών η οποία θα δημοσιοποιηθεί, αν καλά έχω καταλάβει, περίπου τον Οκτώβριο. Και Εντάξει, μπορεί να μην θέλουμε να περιμένουμε την έκθεση της Επιτροπής, άντε να το καταλάβω, αλλά δεν θα έπρεπε τουλάχιστον να περιμένουμε τη δημοσιοποίηση της έκθεσης την οποία παρήγγειλε το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή τον Οκτώβριο. Εγώ θέλω τα πράγματα να γίνονται με τρόπο ξεκάθαρο. Και φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι θα συμφωνούν σε αυτό που λέω. νομοθετώντας πρέπει να λαμβάνουμε τις απόψεις, πρέπει να λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας με τρόπο σαφή. Και να μην κάνουμε τελικά μη ρεαλιστικές προτάσεις. Ξεκινάμε τη συζήτηση από το ESRB και μετά περνάμε σε, στις υπόλοιπες ρυθμιστικές αρχές και τελικά στο, στο ενιαίο σύστημα ρυθμιστικών αρχών. Δεν πρέπει όμως να θέσουμε σε κίνδυνο τις ρυθμίσεις και τις συμφωνίες που έγιναν και με, το, με τη δικιά μας συμμετοχή για παράδειγμα, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πρέπει να συνεχίσει να είναι ε, ε, ο ίδιος και σημαντικός στον τρόπο λειτουργίας της EBA. Δεν πρέπει να έχουμε κάποιο, κάποιο πιστοχώρηση σε αυτό το τομέα. Άρα, κατά την άποψή μου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έπρεπε να προσπαθήσει περισσότερο να βελτιώσει τα πράγματα εκεί που χρειάζεται ξεκινώντας από την υφιστάμενη σημερινή κατάσταση. Δεύτερο θέμα. Υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ της ρύθμισης των τραπεζών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αφενός και των ασφαλιστικών αφετέρου. Πρέπει λοιπόν αυτό να το λάβουμε υπόψη μας στην πρακτική, την καθημερινή λειτουργία αυτής της ρυθμιστικής αρχής. Άρα, ο τρόπος λειτουργίας ή τρόπος ε, λήψης αποφάσεων, ψηφοφορίας ε, θα πρέπει να είναι διαφορετικός. αναγνωρίζοντας τις διαφορές σε καθέναν από τους τομείς. Λοιπόν, τρίτη μου παρατήρηση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να απλοστεύσουμε τα πράγματα οπουδήποτε γίνεται και όχι να κάνουμε το αντίθετο. Διάβασα με προσοχή τις εκθέσεις που είχα στη διάθεσή μου και εγώ θα ήθελα να συνομιλήσω με τους υπεύθυνου αυτών των ρυθμιστικών, ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχιών, αρχών. Θεωρώ ότι για λόγους όχι θεολογικούς αλλά ρεαλιστικούς πρέπει να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε και να συμφωνήσουμε στους τρόπους με τους οποίους η εποπτεία από αυτές τις ευρωπαϊκές αρχές θα γίνει πιο αποτελεσματική. Και σε αυτό το πλαίσιο θα συνεργαστώ με τους, τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές της ομάδας μου. Ευχαριστώ. Οντουλίν. Λοιπόν, Σάντσες, εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Προσωπικά πιστεύω ότι ε, σε αυτή την πρώτη αναθεώρηση θα πρέπει να κάνουμε ένα τσεκ, ένα έλεγχο λειτουργίας των αρχών αυτών στην πρώτη περίοδο και να απαντήσουμε στο ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στη ρήτρα των διαφόρων ε, ε, κανονισμών. Αυτό είναι μια άσκηση που πρέπει να κάνουμε. Υπάρχουν όμως και άλλα θέματα σημαντικά που πρέπει να μας απασχολήσουν. Παράδειγμα, η σχέση με το ε, νέο σύστημα εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενιαίο σύστημα που δεν υπήρχε στο παρελθόν, επίσης τα δημοσιονομικά ζητήματα και τα ζητήματα των πόρων ε, των αρχών αυτών, Κάτι άλλο που θα μπορούσε να μας απασχολήσει είναι πώς να βελτιώσουμε την οικονομική διακυβέρνηση, τη χρηματοοικονομική, εγκρίνουμε πολλά στοιχεία που ρυθμίζουν διάφορα ζητήματα, αλλά θα πρέπει οι ευρωπαϊκές αρχές να ε, συνεισφέρουν ε, σε αυτή την προσπάθεια και την εξέλιξη για το μέλλον. Τώρα, ως προς τον κανονισμό προσωπικά, συμφωνώ να έχουμε ένα κείμενο για τεχνική διαβούλευση ε, και ερωτηματολόγιο ακόμα, δεν ξέρω, εισηγητής να το στείλει στις διάφορες αρχές και να τους δώσουμε και ένα διάστημα να αντιδράσουν για τη διαβούλευση όλα αυτά και για να μπορέσουμε να εργαστούμε καλύτερα. Ως προς τον κανονισμό και τα πιο σημαντικά στοιχεία που θα πρέπει να μας απασχολήσουν, να δούμε αν υπήρξε καμιά δραστηριότητα ε, διαμεσολάβησης. Είδαμε στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της κρίσης ότι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ήταν σχεδόν απούσα τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για το μέλλον και τι βελτιώσεις μπορούμε να προτείνουμε σε αυτό το στοιχείο. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία τραπεζική αρχή διαφορετική από την ΕΜΠΑ και πώς λειτουργούν τα συλλογικά σώματα, πώς λειτουργούν τα συμβούλια, πώς λειτουργούν τα τεστ κοπόσεως. Όλα αυτά είναι θέματα που μας ανησυχούν και είναι και καθημερινή δουλειά τους κανονικά. Ο ε, νέος ε, μηχανισμός εποπτείας είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει ψηφοφορία εκεί, ανάλογα με το ε, αν κανείς συμμετέχει στον ενιαίο μηχανισμό. Και εμείς από πλευρά Κοινοβουλίου θα πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Τώρα θα γίνει ένας έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, λέει. Αυτό θα γίνει σε όλες τις τράπεζες. Έχει λόγο η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Θα ήταν ενδιαφέρον για να είναι πλήρης η διαφάνεια και να μην υπάρχει ε, ανισότητα στους κανόνες παιχνιδιού. Είναι πρακτικά στοιχεία αυτά, αλλά σημαντικά για μένα. Ε, το θέμα του προϋπολογισμού είναι επίσης, μπορεί να έχουν μια αυτονομία, ε, οικονομική που πρέπει να εξασφαλίζεται και στα πλαίσια της ανεξαρτησίας και σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων πάλι μπορούμε να κάνουμε προσπάθειες να προχωρήσουμε να τα βελτιώσουμε πέρα από τη ρύθμιση και χρειάζονται και κίνητρα. Και καλό θα ήταν και ενδιαφέρον να εργαστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και σε ό,τι αφορά τις μελλοντικές συζητήσεις ε, να αναλύσουμε ε, την απόφαση του δικαστηρίου που επίκειται να δούμε κατά πόσον οι εξουσίες των ε, αρχών αυτών μπορούν να μεταφραστούν σε ένα οργανισμό. Δεν ξέρω, πρέπει να βρούμε τη νομική εκείνη ε, μορφή και δομή που είναι καλύτερη. Πώς θα γίνεται η διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με μηχανισμούς μακροπροληπτικής υποπτίας. Στο Κοινοβούλιο προσωρινά επιλέξαμε αυτό να πάει στην κεντρική τράπεζα. Ε, στις ε, Ηνωμένε Πολιτείες ε, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών αυτό. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει η οικονομική μας διακυβέρνηση και προϊόντος του χρόνου να μας απασχολήσει αυτό το θέμα, πώς θα το μεταξελίξουμε. Αυτά όλα είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν με επικοδομητικό πνεύμα και να πούμε ποια είναι και η μελλοντική ατζέντα ενδεχομένω. Και να τα αφήσουμε ανοιχτό. Ως, ε, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, να δούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το σύστημα. Ευχαριστώ. Wolf. Ο Βολφ Κλίντς, ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη από το Σφέν για την καθυστέρηση, αλλά ήμουν σε άλλη συνεδρίαση. Ε, οι τρεις ε, αυτές εποπτικές αρχές ΕΖΑ ε, έχει έρθει η ώρα να αναθεωρηθούν πραγματικά, έχουμε καθυστερήσει κιόλας, αλλά να προσανατολιστούμε προς τα εξής δύο. Όταν συστήσαμε αυτούς τους οργανισμούς, τι εικόνα είχαμε στο μυαλό μας, τι στόχο, αλλά και με βάση ποια δεδομένα και ποιο υπόβαθρο και τι έχει αλλάξει στο μεταξύ. Και εμένα μου φαίνεται ότι τότε είχαμε και την παγκόσμια οικονομική κρίση που μας ε, επηρέαζε και είπαμε ότι χρειαζόμαστε κεντρικές ε, υπηρεσίες που να φροντίζουν ότι η εσωτερική αγορά θα παραμείνει ε, αποτελεσματική. Και αυτή η τάση, οι τάσεις επανεθνικοποίησης και φυγόκεντρες θα έπρεπε να σταματήσουν για να υπάρχει και ένα στοιχειώδες επίπεδο ας πούμε, ίσων κανόνων παιχνιδιού. Κοιτάζω λοιπόν αυτές τις τρεις εποπτικές αρχές και ε, το πόρισμα για την κάθε μια είναι διαφορετικό. Διότι δεν μας υποστήριξε 100% το Συμβούλιο. Θέλουμε να είναι ισχυρές αυτές οι εποπτικές αρχές που να έχουν πραγματικά τη δυνατότητα και για τις τράπεζες και για τις ασφάλειες πολύ γρήγορα να ασκούν αυτή την ε, εποπτική τους ε, λειτουργία και να μην είναι ένα χαλαρό συντονιστικό ε, όργανο ή μια υπηρεσία που να συνεργάζεται με τις άλλες. Ε, στο μεταξύ λοιπόν, τι συνέβη. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μπει πλέον η εποπτεία και έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Αν δω λοιπόν τις τρεις εποπτικές αρχές Λέω τα εξή. Η ΕΜΠΑ, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, δεν ανέπτυξε το προφίλ που εμείς θα επιθυμούσαμε. Πού οφείλεται αυτό. Εν μέρη στο γεγονός ότι υπάρχει στην ΕΚΤ τώρα ε, το ενιαίο σύστημα εποπτείας και για διάφορους λόγους. Δεν με νοιάζει αυτό για ποιο λόγο. Στην αρχή ήταν λίγο ατυχής η λειτουργία του Τα τεστ δεν έδωσαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. κατέταξαν ως λειτουργικές κάποιες τράπεζες οι οποίες πολύ γρήγορα αποδείχθηκαν περίπου πτωχευμένες και αυτό ήταν λίγο τυχές επαναλαμβάνω ως κίνηση. Η ΑΙΟΠΑ ε, νομίζω ανταποκρίνεται ε, στη λειτουργία και στο ρόλο που της ανατέθηκε σχετικά ε, καλά και παρόλα αυτά πρέπει να πω ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να προβληθεί ως ανεξάρτητος φορέας σε όλα αυτά τα θέματα της φεραγγιότητας 2 και αμερόληπτος. Ε, τρίτη, η ΕΣΜΑ, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, είναι η πιο ισχυρή από τις τρεις. Ε, κέρδισε σε ειδικό βάρος όλο και περισσότερο και ήδη ε, πλέον γίνεται και πολιτικός πρωταγωνιστής περίπου σε αυτά τα δεδομένα και πρέπει να αναρωτηθούμε μήπως προσπαθεί να διευρύνει τα όρια των αρμοδιοτήτων της. Αν σκεφτώ τον κανονισμό ΕΜΙΡ και τη συζήτηση που κάναμε στις αρχές του έτους ε, σχετικά με όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι η ΕΣΜΑ εν μέρη ε, ήθελε να τροποποιήσει με μέτρα επίπεδου 2 τα μέτρα επίπεδου 1 που είναι τα νομοθετικά. Ε, νομίζω λίγο το παρατράβηξε εκεί. Για το μέλλον όμως τώρα τι προτείνω. Επίσης θα πρέπει να βοηθήσουμε και να κοιτάξουμε πώς η ΕΜΠΑ θα διατηρηθεί σε πλήρη λειτουργία δίπλα στο SSM, δηλαδή να μην υπάρχει ε, ένας διαχωρισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε χώρες Ευρωζώνης και χώρες εκτός Ευρωζώνης και η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, η ΕΜΠΑ, πραγματικά ε, να ε, θέτει τους κανόνες και να δουλεύει καλά και επαγγελματικά. Η ΑΙΟΠΑ τώρα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει αντίστοιχα με το SSM να μεταξελιχθεί σε μια θέση εποπτείας για τον κλάδο των ασφαλιών. Να ε, είναι όχι απλώς συντονιστικό όργανο, αλλά να κερδίσει εκεί κάποιο ειδικό βάρος. Όλα αυτά είναι εφικτά άραγε. Όλα αυτά ε, είναι επαρκώς χρηματοδοτούμενα. Θα το δείξει αυτό η εξέλιξη στο μέλλον. Θα τεθεί το ερώτημα αυτό οπωσδήποτε. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι εμείς θα πρέπει να φροντίσουμε στην μετεξέλιξη των τριών αυτών ε, εποπτικών αρχών να ισχύουν ήδη κανόνες και ήδη γνώμονες και να μην έχουμε τρεις οργανισμούς που αρχικά είχαν σχεδιαστεί ως, πώς να το πω, ειδικοί οργανισμοί, ειδικά ιδρύματα για μεμονωμένους τομείς που έπρεπε να δουλεύουν με αντίστοιχους κανόνες και τελικά ε, έχουν αυτονομηθεί και λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Επίσης η διαφάνεια ανάμεσα στην μακροπροληπτική εποπτεία του ESRB του Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου δηλαδή και των τριών ΕΣ δεν μου φαίνεται επαρκής. Δηλαδή δεν ξέρω πώς συνεργάζονται, δεν ξέρω ποια είναι η διαφάνεια και πώς μεταξύ τους συνεργάζονται και πώς ε, αλληλεπιδρούν και αλληλενισχύονται. Η Thank you. Um, Ευχαριστώ. Δύο είναι τα ζητήματα κατ' εμέ. Θα ήθελα να σχολιάσω. Ε, ο Σβέντα έθεσε ήδη Άρα το βασικότερο είναι ποιες, ποιοι είναι οι νομικοί περιορισμοί και η πρόορη γνωμοδότηση που εξεδόθη. Θα το σχολιάσω εν συντομία, αν και δεν το είχα προβλέψει. Υπάρχουν κάποια πρακτικά ζητήματα που ανέκυψαν από την εμπειρία που είχαμε στην τωρινή μα θητεία με τι τρει ευρωπαϊκέ εποπτικέ αρχέ. Ε, προσφέρουμε προ τη θέμενη αξία όντω, ε, διότι αρκετά προώρα ε, εκδίδουμε γνωμοδότηση πρωτού παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτω ή το 2014, αυτό το πούμε στην έκθεσή μα θα γίνει αναθέτηση θεώρηση. Έχουμε και το Σόλτ selling στο Ηνωμένο Βασίλειο τη σχετική υπόθεση και έχουμε και την άποψη του, ε, γενικού, του εισαγγελέα του Αριουπάγου ε, και τον Νοέμβριο θα έχουμε και την δικαστική απόφαση. Υπήρξαν αντικρουόμενα σχόλια μέσα στην έκθεση. Φανταστείτε τις στρατιές δικηγόρων που έχουν σκύψει και ε, έχουν δώσει διαφορετικές ερμηνείες για το ζήτημα. Ε, προκύπτει όμως με σαφήνεια από τη γνωμοδότηση και θα δούμε τι θα γίνει με την επίσημη τελεσίδικη απόφαση ότι πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ οι εθνικές ε, εποπτικές αρχές ε, δεν μπορούν για λόγους ενιαία αγοράς να υπεσκελιστούν από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές. Βλέπετε λοιπόν την νομιμοποίηση των αρμοδιοτήτων για απαγόρευση ή για διαμεσολάβηση που έχουν οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές και ξέρετε τι πιστεύουν τα κράτη-μέλη και ως δεν ξέρει το δικό του κράτος ε, μέλος τι πιστεύει για το θέμα της διαμεσολάβησης. Συγκεκριμένα που τώρα πραγματευόμαστε, συμφωνώ με το Σφεν, δεν είναι ζήτημα πειθαρχία, είναι ζήτημα ε, γερής κρατεάς νομικής βάσης ε, και άρα δεν θέλουμε είτε σε εθνικά δικαστήρια είτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να προσβληθεί ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών δεδομένων των πολυάριθμων νομικών υπηρεσιών των μεγάλων εταιριών. Γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι κρατέα η νομική βάση, ώστε να μην αποφασίσουν οι δικηγόροι για το τι θέλαμε να πούμε και τι εννοούσαμε. Αυτή είναι η προσθέμενη αξία. Εγώ δεν είμαι βεβαίω νομομαθή, αλλά έτσι το κρίνω από την εμπειρία που έχουμε με τη ΣΕΖΑ και του φακέλου που εξετάζουμε. Υπάρχει και ένα άλλο ερωτηματικό που. Ε, απαιτεί γνώσεις εμπειρογνώμονα. Για το ενιαίο εγχειρίδιο για τις ΕΣΑΣ νομίζω ότι σε ορισμένους τομείς χρειαζόμαστε μεγαλύτερη τεχνική πραγματογνωμοσύνη και κυρίως πρόσβαση σε μια ευρύτερη βάση γνώσεων. Παραδείγματος χάρη, ε, MIFID, ε, υπάρχουν πάρα πολλά τεχνικά ζητήματα και μέσα στο κείμενο προτείνουμε να συσταθούν τεχνικές ομάδες σε συνεργασία με την ΕΣΜΑ, κυρίως για την τεχνολογία που χρησιμοποιείται σε χρηματοπιστωτικές αγορές και ζητούμε ευρύτερους ελέγχους θεσμοθετημένους. Ε, δεν μπορούμε να ζητάμε να κάνουν πράγματα οποία δεν μπορούν να φέρουν σε πέρας λόγω ελλείψεων. Για τη MIFID, παραδείγματο χάρη, του ζητήσαμε πάρα πολλά για τις στρατηγικές συναλλαγών, ε, κυρίως όσε βασίζονται στους αλγορίθμους ε, και σε συνεργασία με την ΕΣΜΑ πάλι βλέπουμε ότι ακόμη και σε εθνικό επίπεδο δεν είναι διαθέσιμη η πραγματογνωμοσύνη για να διεκπαιρεωθεί αυτό το ζήτημα. Οπότε για το ζήτημα των ρυθμιστικών τεχνικών προτιμών πρέπει πρώτα να μεριμνήσουμε ότι θα έχουν επαρκή πρόσβαση σε μια διευρυμένη βάση γνώσεων για να μην υπάρχουν κενά. Όταν προσπαθούν λοιπόν να διεκπαιρεώσουν κάτι πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν του λείπει η πραγματογνωμοσύνη. Και τι χρειαζόμαστε μηχανισμό, ώστε να γίνεται εξωτερική ανάθεση, να βρίσκουν εκτός την πραγματογνωμοσύνη διότι σε ορισμένε ε, περιπτώσεις ε, είναι δύσκολο να την έχουν. Ε, και ποιο είναι το βασικότερο πρόβλημα. Η αξιολόγηση αντικτύπου στον ΕΜΗΡ, παραδείγματο χάρη, έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις για την ανάλυση κόστους ωφέλους και την αξιολόγηση αντικτύπου που φαίνεται σε πέρα στο ΕΣΜΑ. Βλέποντας λοιπόν τις εκθέσεις μέχρι του για τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και τα ITS, βλέπουμε πάρα δεν έχουμε κανένα ποσό. Μα πώς γίνεται στην αγορά παραγωγό να γίνεται αξιολόγηση αντικτύπου και να μην έχουμε ποσά. Ε, βλέπουμε λοιπόν ε, ότι στι αξιολογήσει έχουμε ένα κυκλικό τρόπο σκέψης, ε, ο οποίο όμω δεν συνιστά αξιολόγηση αντικτύπου. τι, ακούμε διάφορε επιχειρηματολογίε, και άμα έρθει κάποιο από τη βιομηχανία για να ασκήσουν ειδική πίεση, εγώ του ζητάω τεκμήρια, αυτέ αποδείξεις ε, και οι, οι κανονισμοί λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι στο απειρόβλητο σε σχέση με αυτή την ανάγκη προσκόμιση τεκμηρίων. Και Αυτά τα ζητήματα τα έχουμε και με τι απαιτήσει για την υποβολή αναφορών, για την ανταλλαγή πληροφοριών, για οποιαδήποτε παράγωγα. Δεν αναφέρονται στην αξιολόγηση αντίκτυπου. Έχουμε την πρώτη εναλλακτική λύση και τη δεύτερη. Με την πρώτη, τι είναι. Αναμετατίθεται η ημερομηνία υποβολή αναφορών και η δεύτερη εναλλακτική δεν μετατίθεται. Και στη δεύτερη εναλλακτική λέμε, α ναι, διατηρείται καθεστική ατάξη. Ε, και ε, δεν λύνουμε τα προβλήματα βάσει υποβολής αναφορών ETD, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών. Μα τι είναι αυτά. Ε, πρέπει αμελητή να υποβάλλεται μία αναφορά και να ζητάμε κάτι. Δεν ε, είναι αποτελεσματική η αξιολόγηση αντικτύπου αλλιώ. Χρειαζόμαστε... Ε, ε, Παραστατικά χρειαζόμαστε αποδεικτικά στοιχεία και επίσης ευρεία βάση γνώσεων. Ε, τώρα, α περάσουμε και στι ομάδε των εμπλεκομένων φορέων. Ε, το σχολίασε και ο Σβέν. Είναι πραγματικό το πρόβλημα εδώ. Πολλέ ΕΣΕΣ ε, έχουν πάρα, πάρα πολλού εμπλεκόμενου φορεί. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μία, ε, έναν εξαιρετικά ποικιλόμορφο τομέα, όπω το τραπεζικό. Έχουμε μεγάλε τράπεζε, μικρέ, έχουμε συνεταιρισμού, έχουμε ιδιωτικέ τράπεζε. Άρα Μέριμνά μας είναι πρώτον να διαφυλάξουμε την ποικιλομορφία, να εισακούονται οι φωνές όλων, όχι μόνο ενός τμήματος και όταν έχετε ένα πολύ περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που εμπλέκονται σε ομάδες ε, εμπλεκομένων φορέων, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαφυλαχθεί αυτή η ποικιλομορφία απόψεων και το ειδικό του βάρο να είναι ίσο. Ε, η ποικιλομορφία των παικτών της αγοράς ε, στην προσφο την πλευρά ε, της αγοράς είτε της πώληση έχει ιδιαίτερη σημασία. Πρέπει να πηχείτε αυτό. 30, ε, η άποψη 30 ανθρώπων σίγουρα δεν απηχεί την ποικιλομορφία των αγορών. Θυμηθείτε τι γινόταν με τα πάνελ ΣΥΖΑ. Τότε υπήρχαν πολυάριθμες ειδικέ ομάδες που εξέταζαν κάθε μεμονωμένο ζήτημα και δεν δίναν το feedback σε μια διευρυμένη ομάδα εμπλεκομένων φορέων που είχε συσταθεί. Αυτό θα έπρεπε να κάνουμε ούτω ώστε με εξορροπημένο και κυρίως δίκαιο τρόπο να εξασφαλίσουμε θέσει θα οι φωνές όλων. Επίσης α δούμε και πώς λειτουργούν αυτές οι ομάδες εμπλεκομένων φορέων είναι περίεργο ε, σε ένα μεμονωμένο μέλος να μην μπορεί να κοινοποιήσει το περιεχόμενο των εγγράφων, να ζητήσει γνωμοδότηση πραγματογνωμόνων ε, για το περιεχόμενο των εκθέσεων ε, φυσικά. Και αυτό δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί αυτή η άποψη είτε την οργάνωσή τους είτε το βιομηχανικό τομέα που εκπροσωπούν. αλλά δεν μπορεί να μην έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιήσουν το περιεχόμενο και να έρθουν σε επαφή με οποιονδήποτε εκτός τη ομάδας των εμπλεκομένων φορέων. Οπότε δεν είναι περίεργο αυτό σχέση με την εντολή που έχουν λάβει. Ε, και κάτι άλλο τώρα που ε, ε, με ενδιαφέρει και με απασχολεί και εμένα η στελέχωση των υπηρεσιών. Δεν είναι θέμα δημοσιονομικό μόνο. Ορισμένες φορές οι ΕΣΑΣ χρειάζονται κανόνες γιατί μόλις ε, τους αναθέσαμε νομοθεσία επίπεδου 1. Αυτό τι σημαίνει, ότι πολλαπλασιάζεται ο φόρτος εργασίας τους. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουν μόνιμες οργανικές θέσεις. Ορισμένες φορές χρειάζονται αποσπασμένους παραδείγματο χάρη. Αλλά τι μου κάνει εντύπωση, ότι τρόπον την ε, ζητάμε από τις ΕΣΑΣ να κάνουν αυτά τα πράγματα και έχουν μπει μέσα σε αυτή την περίεργη ευρωπαϊκή ποσόστοση για τους εθνικούς αποσπασμένους και χρειαζόμαστε γρήγορη κρίση, ούτω ώστε να μπορέσουν οι ΕΣΕΣ εγκαίρω να φέρουν σε πέρα στα καθήκοντά του, να μην έχουν κανένα περιορισμό σε σχέση με τον αριθμό των αποσπασμένων εθνικών υπαλλήλων με του οποίου μπορούν να συνεργαστούν. Ε, όσα περισσότερα θέματα του αναθέτουμε, τόσο περισσότερου εμπειρογνώμονε χρειάζονται, ούτω ώστε εγκαίρω να το φέρνουν σε πέρα. Πρέπει επίση ε, ε, εγκαίρω να έχουμε θεσπίσει του κανόνε με τρόπο ώστε να επιτρέψουμε την πλήρη λειτουργία των ΕΣΑΣ, ε, ταχύτατα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε αυτούς τους κανόνες, να αποκολλήσουμε από τις ευρωπαϊκές ποσοστώσεις ε, εσάς, ε, γιατί έχουν και τη δική τους ποσόστοση 25% για εξωτερική ανάθεση. Πρέπει λοιπόν να δούμε τις απαιτήσει για τη στελέχωση, ούτως ώστε οι ΕΣΑΣ ε, αυτά τα σκαμπανεβάσματα στο φόρτο εργασίας να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν, γιατί μιλάμε για τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα και το ενίο εγχειρίδιο και άρα δεν χρειάζεται μόνιμη πάγια επέκταση του προσωπικού τους, αλλά δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης, γιατί κάποιος μίλησε για για αυτή τη δυνατότητα και είπε ναι, αλλά με χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Όχι, για την ε, κανονική λειτουργία του θα πρέπει να βρούμε εμεί τρόπου για να απελευθερωθούν και να έχουν τη δυνατότητα να έχουν εξωτερικού συνεργάτε. Αυτά είναι τα τέσσερα βασικά πρακτικά ζητήματα ε, που ήθελα να θέσω και περιμένω την ε, νομική γνωμοδότηση. Σάρων Μπόλ, έχω και εγώ κάποια σχόλια να κάνω. Θα ήθελε κάποιο άλλο πρωτού. Ε, πάρω εγώ το λόγο, όχι. Very quickly, because we're now a bit up against time. Um, πολύ γρήγορα γιατί μάλλον έχουμε αρχίσει να καθυστερούμε τώρα. Πού βρισκόμαστε. Πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά γιατί αναμένουμε πολλές εκθέσεις. χρόνο, όμω, ας μην ξεχνάμε ότι η ε, ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει τον Ιανουάριο και την, ε, στην Ολομέλεια του Φεβρουάριο. Επομένω, έχουμε χρόνο στο διάθεσή μας για να λάβουμε υπόψη μας όλες αυτές τις εκθέσεις και να τις συμπεριλάβουμε τελικά στα συμπεράσματα που θα έχουμε στην τελική έκθεση. Τώρα, του ούτου λεφθέντος και προσπαθώντας να προχωρήσουμε βηματικά και προσεκτικά, δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε ποιο ήταν το, το γενικό όραμα, η γενική προσέγγιση αυτής της Επιτροπής ε, για το που μας, την οποία την έδωσε και η έκθεση la Δηλαδή, το γεγονό ότι το εποπτικό Συμβούλιο βρίσκεται τώρα σε μια υβριδική κατάσταση όπου ταυτόχρονα λειτουργεί σαν διακυβερνητικό όργανο και Ενώ ταυτόχρονα οι ρυθμιστικέ αρχές θεωρούν ότι οι απόψεις τους, οι θέσει τους είναι σωστές ανεξαρτήτως της πολιτικής ε, κατάστασης, των πολιτικών προτεραιοτήτων. Οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές έχουν στηθεί με το πρότυπο των agencies, των, των, των οργανισμών της Επιτροπής. Θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας ε, το μοντέλο που έχει εφαρμοστεί για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες όπου ο οργανισμός έχει αποκτήσει μια μεγαλύτερη πρωτοβουλία και μια μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων από την ε, Επιτροπή. Εάν μπορέσουμε να απομακρυνθούμε από αυτό το μοντέλο του οργανισμού και ταυτόχρονα να απομακρυνθούμε από το μοντέλο του, της διακυβερνητικής συνεργασίας, ίσως αυτό μας διευκολύνει. Ίσως να μην μπορεί να γίνει αμέσως αυτό, αλλά στο μέλλον θα μπορούσε. Υπάρχουν για παράδειγμα προβλήματα στην στη, ε, γεγονός ότι η SSM δεν έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Συμφωνώ πάντως ότι οι τρεις ρυθμιστικές αρχές βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο εξέλιξης, όπως ελέγχθη η EBA είχε πρόβλημα με τα τεστ ε, κοπόσεως, αλλά αυτό που τελικά συνέβη ήταν ότι οι εκπρόσωποι στην EBA υπονομεύθηκαν από την πίεση των κρατών μελών δεν είχαν τη δυνατότητα να ασκήσουν τις πρωτοβουλίες τους και να αναλάβουν πρωτοβουλία. Στην ΕΣΜΑ από την άλλη βρισκόμαστε σε ένα πιο αρχικό ε, στάδιο. Με αυτόν τον τρόπο είχαν τη δυνατότητα να οριμάσει περισσότερο αυτή η υπηρεσία και να αποκτήσει και μεγαλύτερο, μεγαλύτερη εξουσία. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε η Κέι. Στον αφορά το ζήτημα των εμπειρογνωμών, το γεγονό ότι χρειαζόμαστε εξειδικευμένη γνώση και κάποιε ειδικέ ομάδε. Επίση, συμφωνώ με αυτά που είπατε για το ζήτημα της αξιολόγησης αντικτύπου, αν και αυτό είναι γενικό θέμα για όλες τις αξιολογήσει αντικτύπου που μας έρχονται από την Επιτροπή. Τις περισσότερες φορές είναι περισσότερο ένα πολιτικό κείμενο, μια πολιτική ανάλυση και όχι τόσο απτά χειροπιαστά στοιχεία στατιστικά. Σίγουρα θα μπορούσε να βελτιωθεί η ε, αξιολόγηση αντικτύπου, αλλά το γνωρίζουμε για την εμπορία μας από την ίδια την Επιτροπή, συχνά προσπαθώντας να καταπτίσουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση αντικτύπου, καταλήγουμε σε μια πολιτική δήλωση. Αυτό λοιπόν πρέπει να το εξετάσουμε γενικότερα. Μιας και περιμέναμε τον Σβέν, έχουμε καθυστερήσει λίγο σχέση με το χρόνο διαγραμμά μας Άρα να είσαι σύντομος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, τα διαδικαστικά πολύ σύντομα. Η κυρία Λούλινγκ είπε ότι δεν έχει νόημα να κάνουμε έκθεση εδώ αν ε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα για να τα συμπεριλάβουμε της δίκης. Δύο μελέτες έχουμε αναθέσει μία για τη μικροπροληπτική εποπτεία και για τη μάκρο είναι η άλλη. 5 Νοεμβρίου θα τις έχουμε και οι συνάδελφοι θα έχουν χρόνο μέχρι 25-26 του μηνός να κάνουν τις τροπολογίες τους. Και εγώ ε, ως εισηγητής θα έχω τα συμπεράσματα των μελετών. Ε, νομίζω ότι χρονικά είμαστε εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν κατάλαβα καλά, θέλει να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση, αλλά εμείς θα ψηφίσουμε πριν καταθέσει την πρόταση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ακουστεί και η δική μας φωνή. Άλλωστε αυτό είναι και η έννοια της ε, εκθέσεως πρωτοβουλίας, να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, που το πάει η Οικονομική Επιτροπή. Για την Ολομέλεια θα δούμε. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να τηρήσουμε έτσι το χρονοδιάγραμμα, να συμπεριληφθούν τα δικά μας αποτελέσματα, να γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το πάμε ως Επιτροπή τουλάχιστον και ταυτόχρονα να μην ζητήσουμε αναβολή και πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί δεν εξυπηρετεί την υπόθεση. επί της ουσίας θα είχα να πω πολλά. Η πρόσβαση στα διάφορα στοιχεία και δεδομένα. Και το είπα και προηγουμένως ε, για την επιθαρχία των υπαλλήλων. Μα δεν χρειάζεται εκχώρηση ε, κυριαρχίας εδώ. Τι είναι η πρόσβαση σε στοιχεία. Θα πρέπει ε, αυτές οι υποπτικές αρχές να έχουν τα στοιχεία στη διάθεσή τους που χρειάζονται για το συντονισμό για τον υποπτικό τους ρόλο. Τι θα πει προσβασιμότητα σε στοιχεία. Όταν έχουμε ένα ενιαίο μηχανισμό, είδαμε στην αρχή της λειτουργίας του εποπτικού μηχανισμού ότι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από χίλιες οι τράπεζες εκείνες που δεν είχαν συμπεριλάβει. Δεν ήξεραν καν τον αριθμό των τραπεζών. Έδιναν έναν αριθμό ε, και οι τράπεζες ήταν ε, χίλιες και πλέον περισσότερες. Για να μην μιλήσω για παράγωγα κτλ. Δεν υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία σε διάφορα κράτη-μέλη. Και για θέματα ουσίας και βασικά πώς θα νομοθετήσω εγώ. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό ε, το έργο των υποπτικών αρχών. Απλώς ε, είναι ατελέσφορο ε, εάν δεν τολμούν να ζητήσουν κάποια στοιχεία για λόγους υπαλληλικής πειθαρχία και δεοντολογίας κτλ. Και στα, στις ΕΣΑ υπάρχει μεγάλη δυσφορία και σε άλλα επίπεδα από αυτά που αναφέρατε δεν είναι μόνο ότι δεν συμμετέχουν όλοι, περισσότερο είναι ότι να συμμετέχουν οι ενεχόμενοι, αλλά να έχουν και ποιοτική συνεισφορά αυτές οι ομάδες των stakeholders. Δηλαδή, όχι τι λένε, να λένε κάτι που να έχει νόημα. Θα περιστώ σε αυτά, δεν έχω χρόνο να επεκταθώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για αυτά που πρότειναν και θα το ξαναδούμε. Και από κοινού θα προχωρήσουμε νομίζω στη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε. Ε, τότε θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεση 4 με 5 Νοεμβρίου, 26 Νοεμβρίου καταληκτική για τις τροπολογίες, 16-17 Δεκεμβρίου το ξανασυζητάμε, ψηφοφορία έκον 20-21 Ιανουαρίου ε, και Φεβρου, Φεβρουάριος, δεύτερη σύνοδος Φεβρουαρίου, Ολομέλεια. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Για πάμε τώρα γρήγορα στο σημείο 9, δηλαδή υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο τομέα, στο φορολογικό τομέα. Ο κύριο Κούτας είναι ο εισηγητής. Συγγνώμη σας, τριμώξαμε χρονικά, αλλά παρόλα αυτά πάρτε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ε, προτείνει η διεύρυνση του συστήματος αυτόματης ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις φορολογικές, ε, ευρωπαϊκές φορολογικές αρχές στα πλαίσια σε της εντατικοποιημένης καταπολέμησης της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής, ε, μερίσματα, κεφαλαϊκά κέρδη, όλα τα, όλες οι μορφές όλα θα προσθεθούν στον κατάλογο των κατηγοριών που υπόκεινται σε αυτό το σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω πως αυτό ανοίγει και το δρόμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε να έχει ένα πιο ολοκληρωμένο, το πιο ολοκληρωμένο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών στον κόσμο και τα κράτη-μέλη θα ανταλλάσσουν το μέγιστο αριθμό πληροφοριών ανάμεσά τους, όπως έχουν δεσμευτεί να κάνουν με τη ΣΥΠΑ ε, βάσει της ε, φάκτα της, ε, του τέταρτου νομοθετήματος ε, για την φορολογική συμμόρφωση των αλλοδαπών λογαριασμών. αυτό συνάδει και με το σχέδιο δράση Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι φορολογικέ απάτε, φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, αλλά και με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπω εκφράσαμε στην έκθεση κλέβα για την καταπολέμηση ε, των φορολογικών παραδείσων φοροαποφυγής και φοροδιαφυγή. Η τωρινή πρόταση επίση ε, καλύπτει τα αιτήματα των κρατών μελών για μια ευρωπαϊκή φάκτα ε, και κατόπιν διμερών συμφωνιών που έχουν τα κάποια κράτη-μέλη με τη ΣΥΠΑ, δυνάμει της ΦΑΚΤΑ και είναι σημαντικό να παραμείνουμε σε αυτή τη δυναμική ούτως ώστε σπευσμένα να εγκρίνουμε και να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε τον νέο κανονισμό βάσει του χρονοδιαγράμματο που εισηγεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, επίσης πιστεύω πως ε, θα πρέπει να είμαστε ε, στην πρώτη γραμμή της θέσπης παγκοσμίων προτύπων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Γι' αυτό το λόγο κάνω κάποιες προτάσεις για να βελτιώσουμε το κείμενο σε τέσσερις τομείς. Πρώτον, προετοιμασία των δεδομένων για την αυτόματη ανταλλαγή ε, απαιτείται πλήρης ε, συμμόρφωση με την ε, κείμενη νομοθεσία για την, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 16-25-2011 είναι μια οδηγία του Συμβουλίου εκεί βλέπουμε τη σχετική διάταξη και βάσει των διεθνών εξελίξεων πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη. Μια άλλη ιδέα που είχα είναι ε, να αξιοποιήσουμε τις διμερείς συμφωνίες θα ήταν υποφέλες για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να διαπραγματευόταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μελλοντική συμφωνία με τρίτες χώρες για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών αντί για την τρέχουσα πρακτική των κρατών μελών, δηλαδή να διαπραγματεύονται σε διμερές επίπεδο με τρίτες χώρες. Ε, όμως αυτό δεν επηρεάζει τις υφιστάμενες συμφωνίες, ε, διότι αυτή η διάταξη θα αρχίσει να ισχύει όταν η τρέχουσα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ. Το κεφάλαιο για του πόρου. Ε, για να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή της οδηγίας, τα κράτη-μέλη θα χρειαστεί να κινητοποιήσουν ανθρώπινους, τεχνολογικούς και χρηματοοικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την ε, περιπλοκότητα και το μέγεθος, των όγκων των πληροφοριών για την αυτόματη ανταλλαγή αρχής γενομένης από το 2015. Για τις κυρώσεις πιστεύω ότι βασικός σκοπός της οδηγίας είναι ελάφρυνση της ε, ε, αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στι αρμόδιες εθνικέ αρχέ, το κράτο μέλο ε, θα πρέπει να δεσμεύεται για την επιβολή κυρώσεων με τρόπο ώστε να ε, αποκομίζει τι απαιτούμενε πληροφορίε. Θα ήθελα να ακούσω τώρα του συναδέλφου. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε για το ΕΛΚ. Νίτρα. E, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να πω ότι καλωσορίζω την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την υποστηρίζουμε. Υπάρχει όμως κάτι που μας λυπεί και αυτό είναι ότι το βασικό κίνητρο πίσω από αυτή την απόφαση είναι το γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες έχουν δραστηριοποιηθεί έντονα στον τομέα της, κατα... της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Δεν θα ήταν καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει αναλάβει την πρωτοβουλία χωρίς να περιμένει να ακολουθήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του όγκου των συναλλαγών, του αριθμού των συναλλαγών και της κινητικότητας των συναλλασσομένων, θα πρέπει να καταλάβουμε ε, ότι ε, ε, αυτό δημιουργεί προβλήματα στον ορισμό της ε, φορολογητέας ύλη από τα κράτη-μέλη. Γνωρίζουμε ότι πολλά κράτη-μέλη δυσκολεύονται όλο και περισσότερο στη διαχείριση του δικού τους εγχώριου φορολογικού συστήματος, ιδιαίτερα όσον αφορά τους άμεσους φόρους. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης αυτή τη στιγμή προσπαθούν να υλοποιήσουν την οδηγία του 2011. Ε, δεν υπάρχει εμφιβολία ότι αυτή η νέα πρόταση θα ενισχύσει την ενιαία αγορά γιατί θα ενισχύσει την, την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, φορολογικών αρχών και αυτό θα βελτιώσει την προβλεψιμότητα του φορολογικού περιβάλλοντος και θα υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία. Σίγουρα επίσης θα ενισχύσει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Τώρα σε σχέση με τις συγκεκριμένες τροπολογίες, πιστεύω ότι ε, η αύξηση του αριθμού των πληροφοριών που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, που θα πρέπει να ανταλλάσσονται, για παράδειγμα τα μερίσματα, είναι καλό. Είναι καλή ιδέα. Αυτό θα βοηθήσει τις φορολογικές αρχές να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα και ήθε αυτό το σύστημα να καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνώ με την πλειονότητα των ε, τροπολογιών που προτείνει ο κ. Γκούτας, ιδιαίτερα ε, την τροπολογία 8, γιατί αυτή δίνει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνάψει συμφωνίες, να διαπραγματευτεί συμφωνίες με τρίτες χώρες. Και Πιστεύω ότι αυτές οι συμφωνίες ε, είναι προ όφελό μα γιατί έτσι θα μπορέσουμε να, έχουμε κοινά πρότυπα σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά. Στο νέο άρθρο 3α ε, ορίζονται κάποιες νέες κατηγορίες πληροφοριών και νομίζω εδώ χρειαζόταν μια διευκρινιστική υπάρχει μάλλον μια διευκρινιστική πρόταση η οποία ίσως δημιουργήσει προβλήματα στην εφαρμογή. Γνωρίζω ότι σε ορισμένα νομικά συστήματα κρατών μελών δεν υπάρχουν ορισμένες από αυτές τις κατηγορίες που αναφέρονται όπως ε, για παράδειγμα τα αποτελέσματα του ισολογισμού. Άρα θα ε, ήταν καλύτερο να υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για τις ε, πληροφορίε που θα απαιτείται να ανταλλάσσουν τα κράτη-μέλη, γιατί ίσω υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί από κράτο σε κράτος. Για παράδειγμα, ε, συνομίλησα με τις ε, πολωνικές φορολογικές αρχές και μου είπαν ότι αυτή η ημερομηνία εφαρμογή που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσω να είναι υπερβολικά φιλόδοξη, ίσω, να είναι υπερβολικά Ε, Ίσως λοιπόν θα πρέπει να το δούμε αυτό για να μην γίνει μια αποτελεσματική η προσπάθεια εφαρμογή αυτής τη οδηγία και θα συνεργαστώ με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Όλε Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγγνώμη κύριε τον Ρομπέρ Χαιρόμαστε πάντα να βλέπουμε ένα παλιό συνάδελφο και το του δώσω καλό καρδό. Καλώς ορίζουμε την έκθεση του κύριου Κούτας. Συμφωνώ με τον κύριο Νίτρας. Νομίζω θα είχε βελτιωθεί η κατάσταση και θα βοηθούσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη αδράσει. Σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείες Ε, μπορούμε να το κάνουμε, αλλά ε, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ε, ευρωπαϊκό εγχείρημα και μετά από τον κύριο Σνόουντεν. Το φάκτα, δεν μπορούμε να το ονομάσουμε EU φάκτα, δεν θα ήταν σκόπιμο κάτι τέτοιο. Ε, επίσης, χρειαζόμαστε ευρεία συνένεση εδώ Το ξέρω ότι είναι ευαίσθητο το θέμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Αλλά δεν θα πρέπει να δίνουμε την εντύπωση ότι το κοινοβούλιο μας έχει ε, μεγάλο κύρος ή μεγάλο λόγο ε, για ε, τα φορολογικά. Ξέρω, όταν γυρνώ εγώ στην πατρίδα μου, μου λένε προς Θεού μην αναφερθεί στη φορολογία. Ε, εντάξει, το ξέρω ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία, αλλά το θέμα είναι τόσο ε, καυτό, τόσο λεπτό, ε, που θα πρέπει να το προσέξουμε. Ο κύριος Γκίγκολτ και άλλοι ξεκίνησαν μια συζήτηση, αλλά αυτή η συζήτηση έρχεται από το 90, θυμάστε, για το φόρο Τόμπιν και τα λοιπά. Και τώρα βρισκόμαστε εδώ που είμαστε και η φορολογική παράδειση. Ξέρετε, εγώ συμμετείχα στην Επιτροπή Κρίμα, αυτή την ειδική επιτροπή, την έκτακτη, ε, που ε, καταργήσαμε το ε, τραπεζικό απόρριτο. Εγώ το καταψήφισα βέβαια. Και έχει πάρει πολύ πολιτική χρειά αυτή η συζήτηση περιφόρων σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Τα θέματα όμω είναι λεπτά και θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτή την ισορροπία πάντα. Ελπίζω να έχουμε και ένα σύστημα, πώς να το πω, που αν μη τι άλλο είναι συγκρίσιμο, εν πάση περιπτώσει, στα διάφορα κράτη-μέλη. Υπάρχουν κάποιες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι πολύ αποτελεσματικά προς ψυχολογία και γνωρίζω τουλάχιστον μία τέτοια χώρα και άλλε χώρε λιγότερο αποτελεσματικέ. Και η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να είναι σε ίδιο επίπεδο παντού, έτσι δεν είπαμε για τους πολίτες αν μη τι άλλο. Τροπολογίες θα κάνουμε σίγουρα, αλλά πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει τελικά πρόβλημα να συμφωνήσουμε. Τελικά όμως όταν ψηφίσουμε, σας συγκετεύω να έχουμε μια ισόρροπη προσέγγιση και να μην θεωρούμε ότι αναλαμβάνουμε κάποια ευθύνη ε, την οποία δεν έχουμε που είναι των κρατών μελών. Και γιατί τη χώρα μου πολύ σημαντική προστασία των δεδομένων, αν δούμε και τις τελευταίες εξέλιξεις των τελευταίων μηνών. Πάντως θα τα βρούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you for the greens. Ε. Ευχαριστώ από τους ε, πρασίνους ο Ρουίτα Βάρης. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω με κάτι που είπε ο Λεσμή, ο συναδελφός μας. Έλεγε λοιπόν ότι στη Σουηδία του λένε μη μιλάς για αυτό το ευαίσθητο θέμα, τους φόρους. Εγώ έρχομαι πάλι από μια χώρα όπου υπάρχει η Τρόικα και το αντίθετο μου λένε. Και για δικαίως. Στην Πορτογαλία ανάμεσα στην ελληνική και την πορτογαλική διάσωση Είδαμε 68 δις ε, μεταφορές πιστώσεων ε, και αυτό αντιστοιχεί στο μνημόνιο ε, της Πορτογαλίας. Οι 20 μεγαλύτερες πορτογαλικές επιχειρήσεις άλλαξαν την έδρα τους με εικονικό τρόπο και μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία και κάνουν στην Ολλανδία ε, τις αλλοδαπές ε, ξένες επενδύσεις. 30 ε, ε, δις ε, επενδύουν στην Ολλανδία αυτό από την αρχή της ε, κρίσης. Ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό απομυζεί την Πορτογαλία από τα έσοδα της. Όλα αυτά πολύ καλά είναι γιατί επενδύεται στην πραγματική οικονομία αλλά στην πραγματική οικονομία της Ολλανδίας όχι της Πορτογαλίας. Καλό θα ήταν να επιστρέφουν οι αποδόσεις των Ολλανδικών επενδύσεων στην Πορτογαλία. Δεν είναι ίδια περίπτωση με την ανακύκλωση χρημάτων που γινόταν ανάμεσα στην Κύπρο και την Ρωσία. Ε, κάτι που απασχολεί πάρα πολύ πολλούς εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο αλλά και τις πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πώς ε, τα σχέδια ε, διάσωσης, συγκεκριμένα το ε, πορτογαλικό σχέδιο διάσωσης, ε, δεν έχει ως αποτέλεσμα τελικά να είναι φερέγγιο το κράτος. Ούτως ή άλλως, πέρα από τα σύνορα θα πρέπει να φροντίζουμε να καταβάλλονται οι φόροι γιατί για οποιασδήποτε συναλλογές θα Υποστηρίζουμε, εξυπακούεται όχι μόνο την αρχή πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και τι προτάσει που κάνει ο συγητή μα, ο κ. Κούτα. Κάποιε ε, χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αλλάξουν. Δεν μιλάμε φυσικά ακόμη για φορολογική εναρμόνιση ε, υπό τη στενή έννοια του όρου. Ε, σίγουρα θα πρέπει να επιτρέψουμε μια μικρή απόκληση ανάμεσα στους φορολογικούς συντελεστές ε, μιλάμε για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, ωραία, αλλά όταν αποκλίνουν υπερβολικά οι φορολογικοί συντελεστές δεν βλέπω σε τι θα μας βοηθήσει. Τέλος πάντων, ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση σε κάθε περίπτωση και ξαναλέω υποστηρίζουμε και την πρόταση της Επιτροπής και τις προτάσεις του κ. Κούτας. Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο και άλλες τέτοιες χώρες θα έπρεπε να αναθεωρήσουν τα φορολογικά τους καθεστώτα διότι προστατεύουν τους κανόνες περί, τραπε, το τραπεζικό απόρριτο παρόλα όσα συμβαίνουν χρειαζόμαστε κοινοτικοποίηση ε, κάποιων τομέων όπως ο φορολογικός κυρίως ε, ε, η φορολόγηση των κερδών είναι κάτι που πρέπει να μα απασχολεί σε δεδομένε κατάστασεις και γι' αυτό θα υποστηρίξουμε του συναδέλφους και θα καταθέσουμε και νέε τροπολογίες ούτω ώστε να ενισχύσουμε το σκέλο που σχετίζεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ζητώ συγγνώμη που μακρηγόρησα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούτο και ευχαριστώ Πρόεδρε για την υπομονή σα. Πρόεδρο, έχουμε ακρόαση, ξέρετε, σε λίγη ώρα, οπότε σύντομα παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι η πρόταση που συζητούμε του κυρίου Κούτας ε, είναι κάτι με το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε σε γενικές γραμμές. Είναι πολύ σημαντική η πάταξη της φοροδιαφυγής και η καταπολέμηση της. Προφανής δεν υποστηρίζει κανείς ε, τη φοροδιαφυγή ούτε τις ε, αξιόπινες πράξεις σχετικά. Ε, και πολλές φορές είναι πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής από την ίδια την αύξηση των φόρων. προφανώς. Γιατί είναι και ένας φαύλος κύκλος. Όσο αυξάνεις τους φόρους θα αυξάνεται και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή. Δεν έχω να προσθέσω πολλά στην πρόταση. Θα κάνω κάποιες προτάσεις ε, που θα βοηθήσουν τον ε, εισηγητή να βελτιώσει την πρότασή του και να ε, προχωρήσουμε συνενετικά. Δεν είναι διαφωνίες, δηλαδή οι τροπολογίες. Την περασμένη εβδομάδα στην Τσεχική Δημοκρατία συνάντησα τη διευθύντρια της ανώτατης φορολογικής αρχής της χώρας μου και εκπροσώπους του Υπουργείου Οικονομικών που ασχολούνται κυρίως με την πάταξη της φοροδιαφυγής και είδαμε το εξής πρόβλημα. Στα δύο κράτη-μέλη της Ένωσης με τα οποία συνορεύει η Τσεχική Δημοκρατία παράγουν ένα καύσιμο ε, που είναι αντίστοιχο με το ε, πετρέλαιο κίνησης, ε, το οποίο όμως δεν είναι τυποποιημένο και δεν εντάσσεται στο ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου. Λοιπόν, η παραγωγοί το δήλωσαν όχι ως καύσιμο, αλλά ως ενεργειακό προϊόν γενικώς χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς είναι και δεν μπορεί να ε, ε ταξινομηθεί στην κατηγορία για να πληρώνει το βονιδικό φόρο κατανάλωση επί των καυσίμων. Το συζήτησα λοιπόν αυτό το θέμα με τις φορολογικές αρχές ε, για να δούμε πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώς θα το χειριστεί η ίδια. Θα γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει όλο και περισσότερες εξουσίες σε αυτά τα θέματα στα δικά της χέρια. Και έχουμε αρκετές αποδείξεις ότι δεν είναι πάντα ο καλύτερος συνομιλητής, ο πιο ανοιχτό και πιο διαφανής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν αυτό το καύσιμο να ταξινομηθεί ως καύσιμο, να μπει στο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να το κάνει αυτό. Και παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην σφετερίζεται τέτοιες εξουσίες, να ψάχνει λύσεις σε κοινοτικό επίπεδο, ναι, αλλά ξέρω ότι αυτά τα ζητήματα της φοροδιαφυγής δεν είναι αντικείμενο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ξέρω ότι είναι ένα ειδικό παράδειγμα, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες που συζητούμε αυτή την έκθεση για να το θέσω υπόψη σας. Είναι σοβαρό, είναι μεγάλη φοροδιαφυγή, χάνει έσοδα το κράτος και είναι δύσκολο να επιληθεί βέβαια μέσα από την έκθεση αυτή. Απλώς ήθελα να το θέσω υπόψη σας γιατί είναι πολύ σοβαρό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στρέτσεκ. Ο κύριος Χουντής παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, άκουσα ότι είμαστε σε πίωση χρόνου και επομένως θα είμαι σύντομος. Άλλωστε αγαπητοί συνάδελφοι η βασική μου παρατήρηση είναι μία, μπορώ να πω και δύο κουβέντες παραπάνω, ότι ενώ δεν συζητάμε για πρώτη φορά το θέμα των φοροαπαλλαγών, της φοροαπάτης, της φοροδιαφυγής. Είναι και πάλι άλλη μια φορά που συζητάμε οδηγίες που πρόσφατα τροποποιήθηκαν και που πρέπει πάλι να ξανά τροποποιηθούν. Αυτό Εκτός των άλλων, κατά την άποψή μου, και εκεί είναι η βασική παρατήρηση σε σχέση με την προτινόμενη οδηγία, ευχαριστώ τον συνάδελφο, έχει κάνει προσπάθεια με τις τροπολογίες του, είναι μια απόδειξη, επαναλαμβάνω, ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και έγκαιρα αυτό το φαινόμενο. Και έτσι ερχόμαστε κάθε φορά να τροποποιούμε με καθυστέρηση και με ελλείψεις τι σχετική, τις, σχετικές οδηγίες και τα μέτρα που έχουμε να κάνουμε. Πιο αναλυτικά, πρώτον, ουσιαστικά και η καινούρια οδηγία που τροποποιείται δεν απαντάει στο ερώτημα πώς καταμερίζεται αυτή η φοροδιαφυγή, η φοροαπάτη τρισεκατομμυρίων ε, ευρώ. Ποιος τα δημιούργησε. Και η προηγούμενη οδηγία και η σημερινή οδηγία ουσιαστικά στρέφει την αντιμετώπιση της ε, φοροδιαφυγής κυρίως στο μέσο Ευρωπαίο πολίτη, που όπως είπε ο συνάδελφος από την Πορτογαλία αλλά συμβαίνει και αλλού, που σήμερα σε συνθήκες κρίσης έχει περικοπές των μισθών και ταυτόχρονα είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία ότι δεν πληρώνει τους φόρους, ενώ ταυτόχρονα προστίθενται και νέοι φόροι. Επομένως δεν αντιμετωπίζει και η καινούρια οδηγία την αιτία του προβλήματος. Επίσης παρά τα βήματα που γίνονται, το αντικείμενο και το πεδίο ε, εφαρμογής δεν περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις, μιλάω βεβαίως για την ανταλλαγή πληροφοριών, για το ΦΠΑ, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τρίτη παρατήρηση είπα ότι θα είμαι σύντομο. Έχει ακόμα ασάφειες στο πώς μπορεί κανείς να ξεφύγει από το να μην δίνει πληροφορίες, παραδείγματος χάρη σε κάποιο σημείο λέει, μπορεί να αρνείται να δώσει πληροφορίες όταν απειλείται η δημόσια τάξη. Ερώτημα προς απάντηση. Κάτω από αυτό τι μπορεί να κρύψει κανείς όσον αφορά την ανταλλαγή των πληροφοριών και βεβαίως αφήνει στο απειρόβητο τους μεγάλους φοροφυγάδες που εκεί γίνεται η μεγάλη φοροαπαλλαγή, φοροδιαφυγή, φοροαπάτη και για, βάζει το όριο και το πεδίο από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Για μας, μια χώρα σαν την Ελλάδα, που βρέθηκε στην κρίση από, όπως αρκετές χώρες το 2008, ένα από τα προβλήματα ήταν ότι με την εκδήλωση της κρίσης έφυγαν κεφάλαια χωρίς να έχουν πληρώσει τους φόρους. Αυτό τώρα θα περάσει απαρατήρητο, δεν θα υπάρχουν πληροφορίες. Γι' αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, θετικά αλλά ανεπαρκή βλέπω τα βήματα, θα κάνουμε σχετικές τροπολογίες. Ε, η γενική μου παρατήρηση που, με την οποία και ξεκίνησα είναι ότι δεν υπάρχει βούληση να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο και ερχόμαστε να, να νομοθετούμε ατελώς και λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, thank you very much. Ε, Ευχαριστώ. Κύριε Κούτας. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ενημερώσω τους συναδέλφους ότι η 1η Οκτωβρίου είναι η καταληκτική για τις τροπολογίες. Η εξέταση των τροπολογιών ε, ε, θα γίνει στις 17 ή 4 με 5 Νοεμβρίου και σίγουρα 4-5 Νοεμβρίου θα ψηφίσουμε στην ΕΚΟΝ, ε, Δεκέμβριο Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ όλους. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Νίτρας, πρέπει να είναι πιο προβλέψιμο το σύστημα. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Σμιτ, είναι λεπτό το ζήτημα και δεν αναφέρθηκα στη ΣΥΠΑ για να προκαλέσω. Ένα παραλληλισμό ήθελα να κάνω. Ε, τα κράτη-μέλη ούτως ή άλλως σε δυνάμει συμφωνίες πρέπει να συμμορφωθούν. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι ακαθόδος το ζήτημα και συμφωνώ μαζί σας για την ευρεία συνένεση που είναι απαραίτητη για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ε, για να απαντήσω στον κύριο Ταβάρε, σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και βοήθειά σας, για τις ε, τροπολογίες ε, που θα καταθέσετε. Είναι ακόμη ένα βήμα στον αγώνα της καταπολέμησης φοροαποφυγής και φορο ε, διαφυγής ε, και ε, συμφωνώ ότι είναι πολύ καλύτερη λύση κατά πολέμηση φοροδιαφυγής παρά η αύξηση της φορολογίας. Κάνουμε μια τέτοια πρόταση. Κύριε Χουντή, καταλαβαίνω πολύ καλά την αποψή σας. Μην ξεχνάτε όμως, όπως είπα ήδη, ότι κάνουμε ένα βήμα παρόλα αυτά. και ενέχει προστιθέμενη αξία το μέτρο αυτό στον αγώνα κατά της ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και άρα οφείλουμε να το υποστηρίξουμε. Κλείνοντας να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους, ευελπιστώ να καταλήξουμε συνενετική λύση και κυρίως να υπάρξει συσπήρωση γύρω από αυτό το δύσκολο ζήτημα. Πρόεδρος, ευχαριστούμε, ευχαριστώ και τους συναδέλφους που ήταν σύντομοι και καταφέραμε να ολοκληρώσουμε. Ο Κλάους Ρέγκλινγκ μας περιμένει απ' έξω ήδη, οπότε θα πάω να τον φέρω. Ε, για να αρχίσουμε την ανταλλαγή απόψεων που έχει προβλεφθεί. Okay, so, uh, I'm pleased to... Ωραία. Λοιπόν, καλωσορίζω και πάλι τον Κλάου Ρέγκλινγκ που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής του ESM, ε, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Η ανταλλαγή απόψε είναι φυσική συνέχεια των συζητήσεων που έκανε η ΕΚΟΝ μαζί σας με την ε, ιδιότητα που είχατε τότε στο EFSF. Τέλος πάντων είναι αυτή η ιστορία και συνεχίζονται οι συζητήσεις με το Κοινοβούλιο που έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μεταξύ άλλων έχουμε τις αποφάσεις για τη χρηματοοικονομική αρρωγή έλαβε ο ESM. Αυτό επηρεάζει άμεσα την πρωτογενή και δευτερογενή νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης και την εφαρμογή αυτής ε, στην ΕΕ. Είναι σημαντικό λοιπόν σε τακτική βάση να γίνονται ανταλλαγές με τον πρόεδρο του Eurogroup και πρόεδρο τον κύριο Τζερόμ Ντούσεμπλουμ Ε, και ε, Επίσης, αυτό που θα μας απασχολήσει είναι νέος εποπτικός μηχανισμός. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου επιβεβαίωσε στις ε, σε αυτά που είπε στις 21 Φεβρουαρίου 2012 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι θα υπαχθεί το σύστημα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να είμαστε λοιπόν, ελέγχουμε. Θα σας δώσουμε το λόγο για ένα δεκάλεπτο και μετά ε, οι συνήθεις ε, χρονοθυρίδες, οι πεντάλεπτες για τις ερωταπεντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Παραμένω ε, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Είμαι ο ίδιος. <laughs> παρόλο που, του EFSF, παρόλο που ταυτόχρονα είμαι και διευθυντή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Ε, έχουμε το κοινό προσωπικό, αλλά διαφορετικού ε, ισολογισμού και φυσικά μια πολύ διαφορετική νομική βάση και δομή το οποίο έχει ε, επιπτώσεις στο, στη, στη λογιστική και στη λειτουργία. Αν και θα τελικά ο στόχος είναι πολύ παρόμοιος. Όπως γνωρίζετε το ESM ε, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ιδρύθηκε πριν από ένα χρόνο, ενώ το EFSF, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, είχε δημιουργηθεί πριν τρία χρόνια, έχουμε συνεργαστεί στενά. Ε, η θεσμική δομή του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, είναι διαφορετική ε, από τους συνήθεις μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν δημιουργήθηκε το προσωρινό EFSF, τα 17 κρατημέλη ε, της Ευρωζώνης ε, ακολούθησαν ένα σύστημα εκτός της ε, συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα, σύστημα διακυβερνητικής συνεργασίας, γιατί ήταν το μόνο που θα μπορούσε να επιτρέψει την άμεση λειτουργία του συστήματος. Τα χρήματα του ESM, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, προέρχονται από τους προπολογισμού τους εθνικούς των κρατών μελών και οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας λαμβάνονται με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη. Οι αποφάσεις που αφορούν για παράδειγμα την εκταμείευση ε, δόσεων. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα ε, τα κράτη-μέλη χρειάζεται να ζητήσουν και να λάβουν ε, έγκριση και δημοκρατική νομοποίηση από τα εθνικά τους κοινοβούλια. Αυτός ο, αυτή η δομή σημαίνει ότι η σχέση του ESM με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι ad hoc και ανεπίσημη. Ε, παρόλα αυτά θεωρώ το διάλογο και τη συνεργασία ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σημαντική. Και είναι. Αντιλαμβάνομαι επίση το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη λειτουργία του ESM. Ε, πιο μακροπρόθεσμα θα μπορούσαμε να αναμείνουμε ότι θα αλλάξει η σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και ESM εάν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν να εντάξουν αυτόν τον μηχανισμό στο πλαίσιο λειτουργίας της συνθήκη. Να ε, σας περιγράψω συνοπτικά τη λειτουργία και τις ε, δραστηριότητες του ESM. Τα 17 κράτη-μέλη του ESM έχουν ε, παράσχει ένα καλυφθέν κεφάλαιο της τάξης των 700 δισεκατομμυρίων και 80 δισεκατομμύρια είναι το καταβιβλημένο κεφάλαιο. Αυτό είναι ε, το μεγαλύτερο διαθέσιμο κεφάλαιο ε, από οποιονδήποτε ε, διεθνή χρηματοοικονομικό οργανισμό. Η δανειοδοτική ικανότητα του ΙΟΣΕΜ ανέρχεται στα 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα το EFSF συνεχίζει να διαχειρίζεται τα προγράμματα στήριξης της Ιρλανδίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας. Συνολικά από κοινού αυτοί οι δύο οργανισμοί έχουν δανειοδοτική δικανότητα 700 δισεκατομμύρια. Από το 2011 το EFSF έχει παράσχει 168 ε, και δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια προς την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα ε, και παραμένουν 19,8 δισεκατομμύρια να εκταμιευθούν. Από τον Ιούλιο και μετά το EFSF δεν έχει τη δυνατότητα σύναψης νέων προγραμμάτων και ε, οποιοδήποτε νέο αίτημα οικονομικής βοήθειας περνάει από το ESM. Το ESM αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόγραμμα βοήθειας του ε, χρηματοπιστωτικού τομέα της Ισπανίας. Ε, έχουν ήδη εκταμιευτεί 41,3 ε, δισεκατομμύρια ευρώ και δεν αναμένουμε περισσότερη χρηματοδότηση από εκεί. Επίσης υπάρχει το πρόγραμμα μακροοικονομικής εξυγένσης για την Κύπρο. Μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας τα 4,5 το μισά από τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν εκταμιευθεί. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 450 δισεκατομμύρια παραμένουν ε, στο ESM και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ακόμα, δηλαδή το 90% της δανειοδιωτικής του ικανότητας. Οι δύο ε, αυτοί φορεί, το EFSF και το ESM μαζί, έχουν ε, εκταμιεύσει συνολικά 212 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2011 και μετά. Θεωρώ ότι η στρατηγική που ακολούθησε το ESM είναι η ίδια ή εν πάση περιπτώσει συγκρίσιμη με τη στρατηγική που αξιοποιεί εδώ και πολλές δεκαετίες, που ακολουθεί εδώ και πολλές δεκαετίες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και ποια είναι η βασική ιδέα. Παρέχονται προσωρινά δάνεια σε χώρες ε, οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στις αγορές για να δανειστούν. Αυτό δίνει ε, χρόνο σε μια ε, χώρα να κάνει τις απαιτούμενες προσαρμογές και μεταρρυθμίσεις, ενώ ταυτόχρονα ε, παρέχει χρηματοδότηση της οικονομίας ε, με ένα λογικό κόστος. Όπως είπα λοιπόν, ακολουθούμε το ίδιο μοντέλο που ακολουθεί το, ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εδώ και χρόνια, με τη μορφή δανείων ομολόγων και ε, το επιτόκιο που χρεώνει το ESM είναι ε, το ίδιο με εκείνο που ε, καλείται να πληρώσει στις αγορές. Προσθέτουμε απλώς ένα μικρό ποσό για τα λειτουργικά έξοδα του ESM. Με άλλα λόγια, η οικονομική βοήθεια από το ESM δίνει το χρόνο στις χώρες να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να ξαναβγούν στις αγορές. Θεωρώ ότι το ESM είναι μέρος μιας συνολικής ε, στρατηγικής για το ευρώ η οποία συμπεριλαμβάνει για τα 17 κράτη-μέλη της Ευρωεγωζώνης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όπου χρειάζεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, με, τις, με τα προαπαιτούμενα έχουν σημειωθεί σημαντικές πρόοδοι όσον αφορά την δημοσιονομική εξυγίανση και τις ε, δομικές μεταρρυθμίσεις. για παράδειγμα, το ε, εργατικό κόστος αναμονάδα στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την, την Ελλάδα και την Ισπανία έχει μειωθεί. Ταυτόχρονα έχει μειωθεί το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών σε αυτές τις χώρες. Έχουν εξαλειφθεί ή μειωθεί επίσης τα ελλείμματα στους προϋπολογισμούς. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, εμφανίζει πλέον πρωτογενές πλεόνασμα. Και αυτές οι προσπάθειες χάνουν τις, ε, ε, επικροτούνται από τις αγορές. Η Ιρλανδία και η Πορτογαλία κατάφεραν να επιστρέψουν στις αγορές μετά τα δεκαετή τους ομόλογα σε αποδεκτά επιτόκια και η Ισπανία ε, κατάφερε να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις αγορές. Επομένως είμαι πεπισμένος ότι αυτή η βοήθεια είναι απαραίτητη και εάν δεν είχε δοθεί αυτή η βοήθεια, ίσως ορισμένες χώρες να είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το κοινό νόμισμα. Ποιο είναι όμως, ποιος είναι ο αντίκτυπος όμως στην πραγματική οικονομία. ο λαός της δικαιούχη χώρες δεν έχει δει ακόμα τα αποτελέσματα και την πρόοδο. Ε, γνωρίζουμε πολύ καλά το πόσο δύσκολα είναι τα προγράμματα προσαρμογής που έχουν επιβληθεί στις χώρες αυτές, την ανεργία και τις περικοπές. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι μόνο πότε αυτές οι προσπάθειες θα επικροτηθούν από τις αγορές, αλλά από πότε θα έχουμε πάλι ανάπτυξη και ε, θα αυξηθεί η απασχόληση. Η εμπειρία από το Διεθνές Νομισματικό Τομείο δείχνει ότι τέτοιου είδους δομικές μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οδηγούν τελικά σε αύξηση της αποτελεσματικότητας και σε ανάπτυξη, αλλά αυτό καθυστερεί. Το δεύτερο εξάμεινο του, της, του τρέχοντος έτους είδαμε κάποια ενθαρρυντικά σημάδια. Έχει μειωθεί η ανεργία, ή μάλλον έχει σταθεροποιηθεί η ανεργία σε ορισμένες ε, χώρες δικαιούχους. Στην Πορτογαλία είχαμε για ε, πρώτη φορά εδώ και δυόμιση χρόνια ε, ανάπτυξη της τάξης του 1,1% που είναι μεγαλύτερη σε όλες, από όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αυξήθηκαν επίσης οι εξαγωγές της Ισπανίας και στην Ελλάδα η κατάσταση σταθεροποιείται. Πιστεύω ότι η Ευρωζώνη συνολικά βελτιώνει την οικονομική της διακυβέρνηση. Είχαμε την πρώτη και τη δεύτερη δέσμη οικονομικής διακυβέρνησης, ε, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, στοιχεία τα οποία ε, έχουν αναγνωριστεί από τους αγαγορές ως σημαντικά Το ερώτημα όμως πάντα παραμένει αν αυτοί οι κανόνες οι οποίοι υιοθετούνται τελικά θα εφαρμόζονται στην πράξη. Ένα άλλο στοιχείο που παρακολουθούν στενά οι αγορές είναι η Τραπεζική Ένωση. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η τριμερής διάλογος για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Και υπάρχουν και άλλα στοιχεία που θα είναι απαραίτητα για να φτάσουμε στην Τραπεζική Ένωση. Ο ESM είναι ένα μικρό λιθαράκι σε αυτήν την Τραπεζική Ένωση. Όπως γνωρίζετε, οι Υπουργοί Οικονομικών πριν από λίγους μήνες συμφώνησαν στα κύρια στοιχεία αυτής της Τραπεζικής Ένωσης, την οδηγία για την εξηγήση των πιστοτικών ιδρυμάτων το μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης, το οποίο ακόμα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή, θα ε, υλοποιηθεί στην πράξη ε, μετά το φθινόπωρο του 2014 όταν γίνουν σχετικέ συζητήσει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μετά θα αρχίσει να λειτουργεί ο ενίο μηχανισμό. Ε, αυτά είχα μια και ο χρόνος είναι περιορισμένο και ευχαριστώ να απαντήσω στις ερωτήσει σα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και μια που είστε εδώ, να σας πω ότι συμφώνησε να δώσει και συνέντευξη στις 12.30 ο κύριος Ρέγκλινγκ μετά ε, τη λήξη συνεδρίασης εκτός εθούσης. Λοιπόν, πέντα λεπτά ε, έρωτα απαντήσεων, Ζαν Πολ Γκουζές από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενική Δευθυντά. θα συνεχίσω από αυτό το τελευταίο που είπατε. Αναφερθήκατε σε συντομία στο Ταμείο Εξυγίανσης των Τραπεζών που ε, σε 10 χρόνια θα είναι πλήρως λειτουργικό. Και τι το ερώτημα, σε αυτή τη δεκαετία ε, ίδρυσης και συλλογή στο Ταμείο, ε, πώς ε, θα γίνεται η εξυγίνηση. Ορισμένοι θεωρούν ότι το backstop θα πρέπει να είναι εθνικό αν κατάλαβα καλά τα όσα είπε χτες ο κύριος Ντράγκη, άλλοι θεωρούν ότι το backstop θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκό, ε, το κεφάλαιο αυτό, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα επέμβει κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περίοδου μέχρι να συγκεντρωθούν ε, τα κονδύλια στο τομέα. Ορίστε, ο Ζαν Πόλα μέσα στο ψητό μπήκε. Θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ κύριε Γκοζές. Έχετε δίκιο. Υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, αλλά παραμένει το ερώτημα τι θα γίνει και μετά τη μεταβατική περίοδο. Αυτή τη στιγμή ε, είναι πλήρως χρηματοδοτημένο το Ταμείο Εξυγίανσης. Παραμένει το ερώτημα αν θα πρέπει ε, να υπάρχει ένα backstop ευρωπαϊκό ή άλλης φύσεως. Αν δούμε τι συνέβη στις Ηνωμένε Πολιτείες, το FDIC που είναι αντίστοιχο ε, σύστημα χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία και έχει και το δικαίωμα να επιβάλλει και περαιτέρω συνεισφορές όταν χρειάζεται. Πάντως είναι ε, αρκετή διευκόλυνση από ε, την Κεντρική Τράπεζα. Έχει χρησιμοποιηθεί δύο φορές μόνο, αλλά είναι καλό να γνωρίζουν οι χρηματοβογορείς ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ε, υπάρχουν και άλλα εργαλεία που χρησιμοποιεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το OMT της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Καμιά φορά είναι καλό να έχεις τα εργαλεία, όχι για να τα χρησιμοποιείς συχνά, αλλά για να τα προβάλλεις και να ξέρουν οι αγορές ότι υπάρχουν και να ε, Το SRM δεν ξέρω πώς ακριβώς θα λειτουργήσει, ε, ο νέος μηχανισμός δηλαδή εξηγήσεις, η ανάγκη για τον backstop υπάρχει λαμβάνω υπόψη μου και σημειώνω τις συζητήσεις που γίνονται. Αναφέρθηκε ο μηχανισμός σταθερότητας, αλλά είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή δεν θα είμαστε σε θέση να εξασφαλίσουμε αυτό το ρόλο. Θα χρειαζόταν αλλαγή στην ίδια τη συνθήκη και στον κανονισμό ε, για τον ΙΣΕΜ. Αυτό χρειάζεται ομοφωνία και των 17 ε, κυβερνήσεων αλλά και των 17 κοινοβουλίων που εκείρωσαν. Ε, Ζωάν, πολύ χρόνο. Θέλεις να επανέλθεις? Όχι. Η Ελίζα Φερέιρα. Α, όχι, όχι, μια, μια μικρή ερώτηση ο κύριος Κούζες. Κύριε Γενικέ, ε, μιλήσατε για τις χώρες που είναι σε προγράμματα. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα επανόδο τους στην αγορά ή στις αγορές. Σε περίπτωση ε, που δεν μπορούν να τηρήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα υπάρχει κανένα αντίστοιχο σχέδιο. Ε, δεν είναι θέμα σχεδίου διάσωσης, αλλά υπάρχει δέσμευση ε, του Eurogroup και γραπτή ε, στα τέλη του περασμένου έτους ότι οι χώρες που χρειάζονται κάποιους ε, όρους και προϋποθέσεις δεν θα φεθούν στη μοίρα τους αν δεν μπορέσουν να επανέλθουν στις αγορές. Βέβαια, ο στόχος κάθε προγράμματος προσαρμογής είναι να επιστρέφουν στις αγορές οι χώρες και να μπορούν να χρηματοδοτούνται μόνοι τους από τις αγορές χωρίς ε, έκτακτη χρηματοδότηση σε λογικά επιτόκια. Τώρα μπορεί να δείτε τις διάφορες χώρες και να έχετε τις απόψεις σας για το πόσο έχουν προχωρήσει. Προφανώς η Ιρλανδία είναι πιο πέρα από την Ελλάδα, αλλά η Ιρλανδία ήταν και η πρώτη χώρα που δανείστηκε από το Ταμείο, το ΙΦΣΕΦ και οι ανάγκες προσαρμογής της Ιρλανδίας ήταν σημαντικά μικρότερες από ό,τι ε, της Ελλάδας. Ξέρετε το πρόγραμμα της Ιρλανδίας τελειώνει τέλη του έτους. Έχουν βγει στις αγορές και έχουν βγάλει και δεκαετία κρατικά ομόλογα σε λογικά επιτόκια. Ε, είναι κάτω του 4% το επιτόκιο για τα δεκαετή ομόλογα, τα κρατικά της Ιρλανδίας. Είναι αποδεκτό επιτόκιο. Δηλαδή είναι σε καλό δρόμο, πολύ καλό η Ιρλανδία ξαναβγεί στις αγορές. Η Πορτογαλία άρχισε, μπήκε στο πρόγραμμα 6 μήνες μετά, Οπότε μοιραία δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο η Ιρλανδία. Είχαν και λίγα περισσότερα πολιτικά προβλήματα τους τελευταίους μήνες που μεταφράστηκε στη δευτερογενή αγορά σε υψηλότερα επιτόκια. Είναι γύρω στο 7%. Δηλαδή απέχει περισσότερο η Ιρλανδία αλλά το πρόγραμμα της Πορτογαλίας έχει ακόμα 9 μήνες. Είναι μέχρι τα μέσα του 2014 και είναι πολύ νωρίς ακόμα να πούμε τι χρειάζεται μετά να γίνει. Βέβαια ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός σταθερότητα έχει μια πλειάδα εργαλείων και μέσων στη διάθεσή του. Αν θέλει να τα χρησιμοποιήσει το Eurogroup μπορεί. Η Ελλάδα είναι η πιο δύσκολη περίπτωση, αλλά το πρόγραμμα τελειώνει τέλη του 2014 στην Ελλάδα και υπάρχει δέσμευση να βοηθηθεί η χώρα. Ξέρω ότι ο κύριος Ντέιζελμπλουμ όταν ήρθε εδώ σας είπε ότι ε, θεωρεί ότι είναι μάλλον πιθανό να χρειαστεί και περαιτέρω βοήθεια μετά το τέλος του δευτέρου προγράμματος και νομίζω αυτή είναι αυτή τη στιγμή η σωστή εκτίμηση. Ευχαριστώ. Και τώρα η Ελίζα Φερέιρα, που είναι και η συγγήτρια για το μηχανισμό εξηγίας. Ευχαριστούμε που ήρθατε ενώπιον μας. Εξεπλάγει θετικά όταν ε, αναφέρατε πως το ταμείο αυτό, ε, συγγνώμη, Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορούσε ενδεχομένως να δημιουργήσει μία γραμμή πίστοσης για το Ταμείο Εξυγίανσης. Ε, θα με ενδιαφέρε να γνωρίζω περισσότερες λεπτομέρειες σε ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να αναλάβει αυτό το ρόλο διότι το backstop, το αποθεματικό είναι καταλητική σημασία κατά τη γνώμη μου. Υπό ποιες προϋποθέσεις λοιπόν θα διενεργηθεί η άμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών που όπως αναφέρθηκε θα είναι δυνατό μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Εποπτείας. Ξαναλέω, οι υποποίες προϋποθέσεις θα μπορέσει στην πράξη ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας να χρηματοδοτήσει μία τράπεζα. Ειδικότερα, Βραχυπρόθεσμα προβλέπεται να ε, προβούμε σε αυτή την balance και asset review αναθεώρηση του ενεργητικού και των ισολογισμών. Ακόμη όμως δεν έχει δημιουργηθεί το Ταμείο Εξυγίανσης. Θα λέγαμε ότι ο μηχανισμός σταθερότητας που έχει αναλάβει τη διαχείριση θα πρέπει να προβλέψει τη χρηματοδότηση των τραπεζών βάση των συμπερασμάτων αυτής της asset review που θα γίνει, σε ποιο μέτρο θα χρειαστεί τα κράτη-μέλη να παράσχουν και εχέγγυα για να υλοποιηθεί αυτό το εγχείρημα. Αυτές τις δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις θα ήθελα να μου απαντήσετε. Απάντηση. Ευχαριστούμε κυρία Φερέιρα. Ε, ίσως υπήρξε πρόβλημα γλωσσικό. Διορθώστε με. Ε, είπαμε ότι ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα ενδεχομένω θα μπορούσε να δημιουργήσει γραμμή πίστοση. Δεν το είπα αυτό. Είπα ότι θα γίνει συζήτηση. Δεν έχουμε τέτοιο εργαλείο. Ε, προϋποθέτει η τροποποίηση τη συνθήκη κάτι τέτοιο και ε, θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη αν θέλουν να ακολουθήσουν αυτή την άγουσα. Για το ειδικότερο ερώτημά σα, δηλαδή πώς ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας θα μπορέσει να παράσχει χρηματοδότηση σε μεμονές ε, τράπεζες στα πλαίσια της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης αυτών. Εκεί έχουμε τη συμφωνία του Eurogroup ε, για τα ειδικά χαρακτηριστικά special features αυτού του οργάνου δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτό θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί και η BBRD για να είναι συμβατές οι διατάξεις, οπότε ε, χρειάζεται ομόφωνη απόφαση των 17 κυβερνήσεων και σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται έγκριση από το Κοινοβούλιο, αλλά θα έχει δημιουργηθεί έτσι το εργαλείο, δεν προϋποθέτει η τροποποίηση συνθήκης, μόνο ομόφωνη απόφαση των 17 ε, μελών της Ευρωζώνης. Αν υποθέσουμε ότι θα δημιουργηθεί, για να το ξεκαθαρίσω δεν υφίσταται ακόμη, Ξέρουμε όμως ποια είναι τα βήματα που θα το επιτρέψουν. Αν τελικά δημιουργηθεί και αντιμετωπίσει προβλήματα μία τράπεζα, έχουμε προβλέψει τη σειρά αποζημίωσης. Μέτοχη πρώτη, ή μάλλον την ε, τη σειρά αυτών που θα συμβάλλουν. Πρώτα οι μέτοχοι και συνέχεια αν δεν χρειάζεται θα διαγραφούν. Στη συνέχεια θα έχουμε τους κανόνες BBRD όταν υπάρξουν και Ε, θα δείτε μετά ε, πότε θα αρχίσουν να ισχύουν οι κανόνες. Ε, πάντως από 1η Αυγούστου του 2014 αρχίζουν να ισχύουν οι κανόνες και χρειάζεται bail-in από τους πιστωτές της τράπεζας. Ε, ακόμη και φτάνουμε μέχρι τους καταθέτες, αν χρειαστεί. Και στη συνέχεια προβλέπεται και θα υπάρξει αυτό το περιθώριο της άμεσης ανακεφαλαιοποίησης. Είναι η έσχατη λύση ε, που προσφέρει ο ESM ε, στο μέτρο που θα δημιουργηθεί το εργαλείο, το τονίζω, πρέπει να περιμένουμε πρώτα απ' όλα την BRRD. Ε, αναθεώρηση ποιότητας ενεργητικού στη συνέχεια και τεστ κοπόσεως. Αυτά θα μας δείξουν ποιες τράπεζες έχουν ε, ε, κενά, ε, κεφαλαιακά κενά. Και άρα θα κρίνουμε πότε απαιτείται ανάληψη δράσης. Ο κύριος Δράγκη εχθές σας είπε νομίζω ότι αναμένεται αυτό στα μέσα του 2014 και τότε δηλαδή θα γνωρίζουμε αν η κατευθυντήρια γραμμή για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση θα είχε εγκριθεί από τις 17 κυβερνήσεις ε, και στο μεταξύ θα έχετε μάλλον συμφωνήσει για την ε, BRRD με το Συμβούλιο και τότε θα μπορέσει να επέμβει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός. Αυτή είναι η χρονική αλληλουχία ε, και σε κάθε περίπτωση είναι η έσχατη λύση, η χρηματοοικονομική συνδρομή των μετόχων και των λοιπών ε, προηγούνται της έσχατης λύσης. Ε, Ελίσα, δεν ξέρω, τώρα δεν έχουμε πολύ χρόνο, ίσως να επανέλθει στη συνέχεια μας περισσέψει χρόνος. Κλίντς. Ευχαριστώ κύριε Ρέγκλινγκ για τα λεγόμενά σας. Πρώτον, Χαίρομαι για την αισιοδοξία σας ε, και με την οποία αντιμετωπίζετε τη δουλειά σας, γιατί χρειάζεται ε, αισιοδοξία στη ζωή. Γιατί η πραγματικότητα ε, μιλάει με άλλη γλώσσα εν μέρη. Οι δύο προλαλήσαντες αναφέρθηκαν σε αυτό το θέμα και ποιος θα είναι ο μελλοντικός ρόλος του οργανισμού σας. Εμείς εργαζόμαστε με την εξυγίαση και για το χρηματοπιστωτικό τομέα ε, ότι θα πρέπει αυτός να αναλαμβάνει και όχι ο φορολογούμενος. Δεν ξέρω αν χρειάζεται τροποποίηση της συνθήκης, ε, αλλά ο ESM θα πρέπει ε, τουλάχιστον προσωρινά να δώσει χρήματα για το SRM, για τον ενίο μηχανισμό εξυγένσης που δεν έχει στηθεί ακόμα, να μην τα πληρώνουν οι φορολογούμενοι τώρα της μιας χώρας υπέρ των φορολογουμένων μιας άλλης χώρας. Ο κύριος Άσμουσεν θα πρέπει να το δει και ως πραγματικότητα και το συζητάει κιόλα ή μάλλον θα πρέπει να το συζητήσουμε ε, και για την ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε από τώρα αλλά δεν μπορούν να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα εάν δεν ξέρουμε πώς θα λυθεί το θέμα, εάν υπάρχουν κάποια προβλήματα και δυναμίες. Χρειάζεται και χωρίς τροποποίηση των συνθήκων να είμαστε σε θέση ε, να προχωρήσουμε. Ε, περίπου συγκρίνατε το ρόλο σας με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Κοιτάξτε, υπάρχει εδώ εξή διαφορά. Το Δούνο του εργάζεται κυρίως με χώρε που έχουν δικό του νόμισμα. Και μπορεί πάντα να χρησιμοποιεί το εργαλείο της υποτίμησης του νομίσματος. Το έχει κάνει επανειλημμένα ε, για προγράμματα μεταρρυθμίσεων. Πάντα, πάντα, παγίως ε, ζητούσε και πετύχανε στη μεταβατική περίοδο υποτίμηση. Εδώ όμως έλα που δεν γίνεται στην ε, Ευρωζώνη Γι' αυτό ε, ε, ένα προς ένα σύγκριση ε, κατά αναλογία δεν είναι σωστή. Και επίσης μιλήσατε αισιόδοξα για όλες τις χώρες και τελικά και για την Ελλάδα. Μόλις είδα μια ανάλυση του Μπρόγκελ που καταλήγει στο εξή. Ακόμα και αν διατηρηθεί το πρωτογενές πλεόνασμα, ακόμα και αν υπάρχει ανάπτυξη, δεν ξέρω, 1,5% τελειώνω. Τα, οι απώλειες θα είναι 170 και με 175% του ΑΕΠ ε, το 2020. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κλίντς. Απάντηση. Στα αγγλικά. Ε, επιτρέψτε μου να σχολιάσω το δικό σας σχόλιο. Ξέρετε ότι ε, συχνά με χαρακτηρίζουν υπεραισιόδοξο. Το έχω συνηθίσει. Όταν παρουσίασα πριν από 15 ε, μήνες ε, την άποψη ότι είμαστε σε καλό δρόμο προς τις αγορές και ότι θα παραμείνει ε, το ευρώ ενωμένο. Μπορεί να υπάρχουν διάφορα στοιχεία κρίσης, αλλά εμείς θα καταφέρουμε να τα ξεπεράσουμε. Ο κόσμος δεν με Νομίζω ότι η τότε μου αισιοδοξία δικαιώθηκε. Ελπίζω να δικαιωθώ ξανά. Είναι πολύ μεγαλύτερη η πρόοδος από ό,τι γενικά ο κόσμος αλλά και τα μέσα ενημέρωσης παραδέχονται. Για το δεύτερο σχόλιο σας έχετε δίκιο. Ε, υπάρχουν ε, όλες αυτές οι διαφορετικές προσπάθειες ε, και στην Τραπεζική Ένωση ποιος είναι ο στόχος ο φορολογούμενος να πληρώνει πολύ λιγότερα στο μέλλον από ό,τι στο παρελθόν. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε. Και το bail-in, η εσωτερική διάσωση, θα πρέπει να επανειδωθεί. Εγώ δεν είπα ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, θα πρέπει να, είναι, να δίνει το απόθεμα, το backstop για το μηχανισμό εξυγίασης. Γι' αυτό χρειάζεται τροποποίηση των συνθήκων. Αλλά σας παρέπεμψα και στην εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκεί υπάρχει σαφής ε, ε, κατάσταση και προηγούμενο ότι δεν χρειάζονται χρήματα από των φορολογουμένων, αλλά να υπάρχει αυτή η δυνατότητα για να καθησυχάζονται οι αγορές, ότι έχουμε ένα πόθεμα, ένα backstop, ε, ε, ένα φρένο ε, και αν υπάρξει αυτό για το SRM δεν θα το πληρώσουν οι φορολογούμενοι αλλά οι ίδιοι οι ενεχομένοι του κλάδου προς το μηχανισμό εξυγίανσης για να υπάρχει εμπιστοσύνη. Θα είναι μια προσωρινή χρηματοδότηση, αλλά όπως σας είπα δεν ξέρω τι ρόλο θα παίξει εδώ ο μηχανισμός σταθερότητας ή αν παίξει καν. Έχετε επίσης δίκιο όταν λέτε ότι χρειάζεται σαφήνεια όταν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των ε, τεστ κοπόσεως και των ε, ε, αναθεωρήσεων των στοιχείων ενεργητικού. Είπατε ότι είναι λάθος η σύγκριση με το δυνατό; Αν μου επιτρέπετε διαφωνώ ε, με την απόψή σας. Πολλά ε, προγράμματα μεν του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χρησιμοποίησαν τη συναλλαγματική ισοτιμία ως μία μεταβλητή ε, προσαρμογής. Προφανώς για το ευρώ αυτό δεν γίνεται. Αλλά τι είδαμε στην Ευρωζώνη την τελευταία τετραετία. Χρησιμοποίησαμε αντίστοιχα ισοδύναμα εργαλεία για να φτάσουμε στον ίδιο στόχο σε χώρες όπως η Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία και προηγουμένως τη Λετωνία που το νόμισμά της συνδέεται με το ευρώ έκαναν ε, περικοπές στα εισοδήματα ε, και τελικά εσωτερική ε, υποτίμηση. Ε, ονομαστικά περικοπές είναι ε, στη Λετωνία, στην ε, Ελλάδα, στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και η ανταγωνιστικότητά τους γρήγορα επανέρχεται. Ισχύει λοιπόν αυτό το θέμα με το δυνητού. Εγώ πρέπει επίσης να πάρω τα χρήματα από τις αγορές, ενώ το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τις κρατικές κεντρικές τράπεζες. πρέπει να σταματήσω. Συγγνώμη, Βόλφο, αλλά μίλησες στην ερώτησή σου και δεν έχεις άλλο χρόνο. Από την ECR η Βίκη. Thank you very much. Ευχαριστώ ε, μας διαφωτίζεται για κάποια πολύ περίπλοκα ζήτηματα. Αν σας κατάλαβα καλά και σβήνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, θα μπορεί να προβλέψει για το Ταμείο Εξυγίανσης το backstop, αλλά με την έγκριση των 17 κυβερνήσεων θα μπορέσετε να κάνετε άμεση ανακεφαλαιοποίηση, αλλά στα πλαίσια επιμερισμού ευθύνης ε, που προβλέπετε στους κανόνες για τις κρατικές προμήθειες και στην PRRD. Ερώτηση λοιπόν. Αν είναι να κάνετε ένα βήμα παραπάνω, τροποποίηση της συνθήκης ε, και να παράσχετε τουλάχιστον ε, μία εγγύηση για το Ταμείο Εξυγίανσης ε, στην περίοδο οικοδόμησής του. τι θα γίνει, πώς θα μεταχειριστούμε μια χώρα που δεν ήταν στους 17 αλλά μετήχε ως ε, κράτος μέλος στο SRM, στον ενίο μηχανισμό. Αυτές οι χώρες δηλαδή που προτίθενται να συμμετάσχουν αλλά δεν είναι στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται με αυτές τις χώρες. Ναι, πολύ σημαντικό το ερώτημά σας, αλλά δεν έχει συζητηθεί σε επίσημα βήματα ακόμη. Ε, προκύπτει όμως ε, επανειλημμένα. Ε, στο άτυπο Εκοφίν στο Βίλνιους πριν από 10, μέρες, 10 μέρες συγγνώμη, προέκυψε. Αλλά δεν έχουμε ξεκαθαριστεί τα πράγματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιδιώξουμε τροποποίηση της συνθήκης ούτως ώστε να χρησιμοποιείται το ταμείο backstop για τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Ακόμη ε, δεν έχουμε σκεφτεί και ένα άλλο επιπρόσθετο δύσκολο ζήτημα τι, πώς να μεταχειριστούμε τις ε, χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωζένα παρόλα αυτά συμμετέχουν στην Τραπεζική Ένωση πρέπει να βρεθεί μια λύση, διότι όπως σας είπα κάνω στον παραλληλισμό με τσίπα, αλλά είναι και λογικό, χρειαζόμαστε με κάποιο τρόπο ένα δημοσιονομικό αποθεματικό. Η έκτεξε καθάρισε ότι ε, αυτή αυτό το επιπρόσθετο καθήκον ενίο επόπτης προϋποθέτει ότι θα έχουμε ένα αποθεματικό όχι μόνο μέχρι να αισθηθεί το Ταμείο αλλά και μακροπρόθεσμα. Δεν ξέρω από που θα προκύψει, είναι ε, το ζήτημα, το, ε, δεν το έχουμε ρυθμίσει αλλά είναι κατεπήγον επίσης. Βίκη, επερώτηση. Χαίρομαι που συμφωνήσαμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο το ζήτημα. Ε, Μπολς, ναι, κάποια πράγματα είναι δύσκολα. Σμεν Γκίγκολ, πράσινη. Ναι κύριε Ρέγκλινγκ, σας ευχαριστώ και πάλι για την επισκεψή σας και επίσης σας ευχαριστώ που απαντήσατε στις γραπτές μας ερωτήσεις. Αυτό βοηθάει και στη δημιουργία εμπιστοσύνης. Είδαμε τα αποτελέσματα σε εκλογές σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες και πιο πρόσφατα στη Γερμανία, παραλίγο να μπει στη Βουλή ένα αντιευρωπαϊκό κόμμα, στην Bundestag. Δόξα το Θεώ, το γλιτώσαμε αυτό το ποτήρι. Και ε, βλέπουμε και στις άλλες ε, χώρες εκλογικές αναμετρήσεις και αποτελέσματα. Και πολλοί πολίτες δεν ε, προβληματίζεται μόνο για την οικονομική και την κοινωνική εξέλιξη, αλλά σου λέει και ποιος έχει το δημοκρατικό έλεγχο. Ε, τα κοινοβούλια ή μήπως χωρούνται και μετατοπίζονται ε, οι αποφάσεις σε κάποια σκοτεινά κέντρα. Ο κύριος Φαναρόμπο μας είπε προηγουμένως στην Ολομέλεια ότι το ESM θα υπόκειται στην αυστηρή στον αυστηρό έλεγχο του Κοινοβουλίου, στις 27 Ιουνίου απαντήσατε σε μια αλληλογραφία εσείς ότι η σχέση σας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν πολύ και να επιβαρύνουν πέρα από την υποχρέωση αναφοράς που έχετε και ότι τα πιο συγκεκριμένα και τα πιο αυστηρά θα τα δούμε αργότερα. Και λόγω των δομών είπατε ad hoc και άτυπα θα πρέπει να ασκούμε τον έλεγχο. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Στο EFSF, στην ιστοσελίδα τουλάχιστον, γινόταν αναφορά στα δικαιώματα του Κοινοβουλίου. Στον ESM αυτή η αναφορά έχει εξαφανιστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εμφανίζεται πουθενά στην ιστοσελίδα του Μηχανισμού Σταθερότητας. Σας ερωτώ, είστε διατεθειμένος τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να τα σεβαστείτε τα δικαιώματα ερωτήσεων, το γεγονός ότι έρχεστε εδώ για ακρόαση, να τα τιμάτε αυτά τα ε, δικαιώματα και να τα υλοποιείτε, να τα διασαφηνίσετε. Εσείς θα δώσετε στο Κοινοβούλιο δικαίωμα συμμετοχής ως παρατηρητή στα όργανά σας. Είστε διατεθειμένος και γραπτά ε, να δεσμευτείτε ότι θα απαντάτε σε ερωτήματα που μας ε, δίνουν ψηφοφόροι μας για σας. Και επίσης γίνεται ουσιαστική συζήτηση στα οργανά σας ή έγινε για το θέμα των δημοκρατικών ελέγχων και δικαιωμάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εντάξει, μπορεί να είναι διοργανική αυτή ε, η συνεργασία, αλλά δεν θέλετε να δώσετε δικαιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διμερώς. Ε, είχατε δεσμευτεί γι' αυτό και χαίρομαι και περιμένουμε χαρά την απάντησή σας. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι το νομικό πλαίσιο είναι σαφές και προσπάθησα να το εξηγήσω στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις. Το ESM όπως και το EFSF δεν είναι ε, θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διαπιστώσαμε όταν άρχισε η οργάνωση του ESM και ετέθη το ζήτημα το ποιος θα ενεργεί το ναρκωτό έλεγχο. Συζητήσαμε το ελεγκτικό συνέδριο και τους ρωτήσαμε εσείς μπορείτε, το ελεγκτικό συνέδριο μπορεί να ασκεί αυτό τον έλεγχο. Τον ενδιαφέρει η πιθανότητα, αλλά αφού το εξετάσανε από νομική άποψη, το συμπέρασμα ήταν ότι δεν ήταν δυνατόν. Και αναγκαστήκαμε να βρούμε μια διαφορετική λύση και ο λόγος για όλα αυτά είναι ότι δεν προβλέπεται αυτό το ESM στην ε, συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως τα δικαιώματα του Κοινοβουλίου δεν καθορίζονται πουθενά. Όπως βλέπετε όμως με προθυμία ήρθα και ευχαρίστως ήταν στις ε, ερωτήσεις σας. Το ίδιο θα πράξω και με γραπτά ερωτήματα Εάν μου τα αποστείλετε θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τα απαντήσουμε. Επίσης σας αποστέλουμε την ετήσια έκθεση ε, και την ε, έκθεση ορκού του ελέγχου, την αποστέλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα με τρόπο ad hoc και ε, ανεπίσημο θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να ξεπεραστούν. Αλλά για να επισημοποιηθεί και να θεσμοθετηθεί αυτή η συνεργασία θα πρέπει να το συζητήσετε με κάποιο πολιτικό όργανο, ε, είτε για παράδειγμα ας πούμε, με τον πρόεδρο του Eurogroup, ο κύριος αλλά εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σχολιάσω. Θα ήσασταν πρόθυμος να τα παρουσιάσετε όλα αυτά και στην ιστοσελίδα σας, πρώτον. Δεύτερον, στα όργανα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας συζητήθηκε αυτή η σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι βγήκε. Um, um, ναι. Η ιστοσελίδα μας ικανοποιεί πολλούς εξαιτία του ότι είναι αρκετά αναλυτική και γιατί όχι να μην εξηγήσουμε καλύτερα την ε, σχέση μας. Αλλά αυτό που θα καταγράφαμε στην ιστοσελίδα είναι αυτό που μόλις σας είπα όσον αφορά τη σχέση του ESM και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε και κάποιο σύνδεσμο ε, στο web stream ε, τη ζωντανή μετάδοση αυτής της συζήτησης. Στι συναντήσεις του ESM πρέπει να σας πω ότι είναι συνήθω για την αντιμετώπιση μια κρίσεω, επομένω το ζήτημα που θέτεται δεν έχει τεθεί. Παρ' όλα αυτά, οι Υπουργοί Οικονομικών το γνωρίζουν, το έχω συζητήσει και με τον κύριο Ντάισελμπλουμ. Γνωρίζει λοιπόν το θέμα, αλλά δεν έχει συζητηθεί. Οι Υπουργοί το γνωρίζουν, απλώς δεν... Ε, και θα πρέπει ε, σε εκείνο το επίπεδο, στο επίπεδο των Υπουργών να συζητηθεί η θεσμοθέτηση των σχέσεων Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε επίσης για τις ε, γραπτές απαντήσεις που αποστήλατε στα ερωτήματα που σας είχαμε υποβάλει πριν τη συνάντηση, πριν την ακρόαση. Η Γκούε δεν εκπροσωπείται. Κάπου θα βρίσκονται αλλού οι εκπρόσωποι. Επομένως το ΕΛΚ. Η κυρία. Η κυρία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κούλ. Σας ευχαριστώ κύριε Ρέκλινγκ για αυτές τις παρατηρήσεις, για την περιγραφή που κάνατε για το ESM ως δυνατότητα, ως μέσο χρηματοδότησης και ε, επίσης σας ευχαριστώ και για τις πληροφορίες για την ε, ανακεφαλαιοποίηση Επίσης είναι πολύ ξεκάθαρο ποιο είναι το πλαίσιο της σημερινής ε, συνθήκης και ε, θα ήθελα να γνωρίζω δεν θα είναι για νομικούς λόγους δυνατόν να συμπεριληφθεί το ESM στη νέα νομοθετική πρόταση για τον ε, ενιαίο μηχανισμό. Και δεύτερη ερώτηση. Την επόμενη χρονιά όσον αφορά την αξιολόγηση στοιχείων ενεργητικού και τα επόμενα βήματα μετά από αυτή την αξιολόγηση, τα οποία ας ε, ελπίσουμε δεν θα χρειαστούν. Αν κοιτάξουμε το ταμείο, το πεδίο εφαρμογή του ήταν πολύ πιο μικρό και σαφές, γιατί αναφέρεται μόνο στην ανακεφαλαιοποίηση. Επομένως χρειάζεται μια, ένα σύνδεσμο με το ESM. Επίσης, για την οδηγία για την εξηγίαση πιστοτικών ιδρυμάτων, PRRD. Προβλέπεται εφαρμογή το 2015 για την GSD 2016, το SRM το 2015. Όλες αυτές οι διαφορετικές ημερομηνίες δεν θα δημιουργήσουν κάποια σύγχυση. Για την πρώτη σας ερώτηση δεν μπορώ εγώ να σας πω τι θα συμπεριλάβετε και τι δεν θα συμπεριλάβετε στα ψηφίσματα και στις εκθέσεις σας, όμως πρέπει να έχετε πλήρη επίγνωση των νομικών και εν τέλει πολιτικών ε, προσκομμάτων ε, για κάποιες ε, υποσυζήτηση ιδέες. Και ήθελα αυτό να το διευκρινίσω για να μην υπάρχουν ψευδεστήσεις. Ε, αυτό οδηγεί σε σύγχυση ε, στις αγορές, ε, δυσκολεύονται όλοι να καταλάβουν τις προθέσεις και την προέλευση κάποιων ιδεών. Όντως έχει δημιουργηθεί σύγχυση για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση και το σχετικό εργαλείο αληθεύει ότι μόλι πάρουμε τελική έγκριση, ε, αυτό είναι λιγότερο σημαντικό διότι έχουμε και του κανόνε για τι κρατικέ προμήθειες Ευρωπαϊκή Επιτροπής που προβλέπουν bail-in διάσωση ιδίων πόρων προτού μπορέσει να γίνει η άμεση ανακεφαλαιοποίηση ε, θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τη διαδικασία, αλλά πάντως όντως υπάρχει σύγκριση στις αγορές για αυτά τα δύο ζητήματα κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ως συνομοθέτες ε, συμμετέχουμε σε αυτές ε, τις διαπραγματεύσεις. Τι θα μας συμβουλεύατε λοιπόν ε, για την εφαρμογή. Απάντηση να, ε, το να καταστήσετε όσο το δυνατόν απλούστερη γίνεται τη διαδικασία. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί και αποκλίνουσε απόψεις ανάλογα με το κράτος μέλος και δύσκολα μπορεί κανείς να συγκεράσει αυτές τις απόψεις πρέπει να δώσετε ικανοποιητικές εξηγήσεις, να γνωρίζουν οι αγορές και οι επενδυτές ε, τι ισχύει. Ε, δεύτερη περίοδος, κυρία Βορτμαν Κόλ. Οπότε, ε, εγώ συνάγω το συμπέρασμα ότι θέλετε να πλησιάσουν οι δύο ημερομηνίε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Ναι. Ε, χνέφει καταφατικά ο, ο μιλητής, ο κύριος Παύλο Ζάλμπα Μπιντεγκιά. Ευχαριστώ κύριε Ρέγκλινγκ που ήρθατε σήμερα ενώπιον μας. Θέλω να αφαιρθώ λίγο στην άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Είπατε ότι την αντιλαμβάνεστε ως ε, σχάτη ε, λύση και καταφυγή. Έχω μια αμφιβολία όμως. Είπατε κάποτε ότι η άμεση ανακεφαλαιοποίηση μιας τράπεζας από το ESM καταναλώνει τριπλάσιο κεφάλαιο από τη βοήθεια σε μια χώρα. Αυτό συμπεριλαμβάνεται σε ένα κείμενό σας. Αυτό που το βρήκατε το τριπλάσιο όμως, πώς βγαίνει αυτός ο υπολογισμός. Δηλαδή, γιατί είναι τριπλάσια ε, η άμεση ανακεφαλοποίηση των τραπεζών από το να δίνατε στη χώρα την ενίσχυση. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Πώς το υπολογίζετε. Έχετε δίκιο. Δεν αναφέρεται στις κατευθύνες γραμμές αυτό, αλλά ε, είναι πληροφόρηση που συλλέξαμε από άτυπες επαφές με οίκους αξιολόγησης. Όπως ξέρετε, ε, ο EFSF πριν από τρία χρόνια και ο ESM πρόσφατα προσπάθησε να πάρει τριπλό α ε, στην αρχή. Ε, είχαμε και από τις τρεις, τους τρεις οίκους Τώρα έχει μειωθεί αυτό γιατί έχουν υποβιβαστεί τα κράτη-μέλη Παρ' όλα αυτά έχουμε τριπλό α ή διπλό α συν ε, και για τον ESM από τους οίκους και αυτό είναι σημαντικό να έχουμε μια ευρύτατη βάση επενδυτών. Ορισμένοι επενδυτές όπως είναι κεντρικές τράπεζες αναδειωμένων αγορών δεν θα δήλωναν προθυμία επένδυσης αν δεν είχαμε τόσο καλό βαθμό. Από αυτές λοιπόν τις επαφές ε, ξέρουμε ότι οι οίκοι αξιολόγηση θεωρούν ότι ε, είναι πιο ε, μεγαλύτερο το ρίσκο να επενδύσεις στις τράπεζες παρά να δίνεις βοήθεια σε χώρες. Και αυτός είναι ένας απλός υπολογισμός που κάνουμε ότι αν ε, δίνεις ρευτότητα ε, σε μια τράπεζα, αυτό έχει τριπλάσει ο κόστος από ότι ε, δάνειο σε μια κυβέρνηση. Είναι ένας γενικός αριθμητικός κανόνας, πρακτικός αυτός. Τα γνωρίζουν οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες και τους έχω ενημερώσει. Και γι' αυτό είναι 60 δισεκατομμύρια η οροφή που αναφέρεται για αυτό το μέσο. Βεβαίως υπάρχουν διάφοροι λόγοι, αλλά ένα σημαντικό είναι ότι αυτά τα 60 δισεκατομμύρια αφορούν ε, επί 380 180 από τα 500 που έχουμε. Και επειδή θέλουμε να διασώσουμε μια δύναμη πυρός για τον αρχικό στόχο του ESM, δηλαδή να δίνουμε μακροοικονομικής προσαρμογής δάνεια στις χώρες, πρέπει να περιορίσουμε το ποσό που ε, αφιερώνεται ή που προβλέπεται για άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πάντως η βάση αυτό είναι οι άτυπες συζητήσεις που είχαμε με τους οίκους αξιολόγησης. Uh, thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Ο Αντολίν Σάτσος, ε, πρεσέντο από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, στα βλέσια και των συνθήκων σας και ε, των προγραμμάτων. Είπατε ότι ο μηχανισμός σταθερότητας δεν είναι ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο. Ναι, εντάξει, δεν είναι κοινοτικό όργανο, αλλά είναι ευρωπαϊκός θεσμός. Ε, εργάζεται στην Ευρωζώνη, καλείται να σταθεροποιεί στην Ευρωζώνη, ε, είναι στην Ευρωπαϊκή και Νομισματική Ένωση και βάσει της παρούς συνθήκες. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ευθύνη να ελέγχει ότι οι οικονομικές πολιτικές είναι προς το κοινό συμφέρον και έχουμε ρόλο και στην οικονομική πολιτική. Ε, πιστεύω εγώ και ε, στον δικό σας οργανισμό. Δεύτερον, Βεβαίως υπάρχει ένα δίχτυ ασφαλείας που χρειάζεται για να ολοκληρωθεί το σύστημα τα κράτη-μέλη που έχουν προβλήματα σταθερότητας ενισχύονται, αλλά και εκείνα που μπορεί να μην έχουν πρόβλημα σταθερότητας, αλλά ο χρηματοπιστωτικός τομέας κινδυνεύει. Και έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα τώρα, η άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και μπορεί να αλλάξει με το άρθρο 19, αλλά υπάρχει κάτι που εσείς θέλετε να βασίζεται σε τροποποίηση των συνθήκων. Ε, δηλαδή, με το άρθρο 19 μπορείτε να δίνετε άμεση βοήθεια ή να ανακεφαλαιοποιείτε τις τράπεζες. Για ποιο λόγο χρειάζεται τροποποίηση των συνθήκων θεωρείτε εσείς. Δεν μπορείτε να βασιστείτε στο άρθρο 19. Και στη συνέχεια η Ισπανία έχει ένα μνημόνιο ε, που τελειώνει φέτος, είναι διετές, τελειώνει αυτόματα ή πρέπει να το ζητήσει η Ισπανική κυβέρνηση και να συμφωνήσουν όλα τα μέλη. Πώς είναι η εκπνοή του μνημονίου. I fully agree with that the ESM is a European institution. Συμφωνώ με αυτά που είπατε, αλλά υπό την νομική έννοια δεν είναι θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εσείς μπορείτε να μου αντιτάξετε ότι επηρεάζει τις σχέσεις μας, αλλά με ρωτήσατε για αυτό το ρόλο του backstop για το ESM. Ε, να μην αποφασιστεί δηλαδή βάσει του άρθρου 19 Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης μα ε, όλες οι νομικές υπηρεσίες μας ε, αποφάσισαν ότι είναι ανέφικτο διότι πόρο απέχει από τους αρχικούς στόχους του ESM και άρα χρειάζεται τροποποίηση της συνθήκης. Αυτή είναι η γνώμη των νομικών υπηρεσιών αλλά όπως είπα και σε προηγούμενες απαντήσεις Άρχισε πρόσφατα η συζήτηση και ακόμη δεν έχει προχωρήσει. Μπορεί άλλοι δικηγόροι να καταλήξουν σε άλλα συμπεράσματα. Προς το παρόν όμως αυτή την ανάλυση έχουμε. Ε, για την ερώτηση για την Ισπανία, 150 δις δέσμευση για την αναδιάρθρωση των τραπεζών. Πέρσι ελήφθη αυτή η απόφαση, όπως μας είπατε, και στο τέλος του τρέχοντος ε, ε, θα λήξει το ε, μνημόνιο ε, και η Ισπανική κυβέρνηση επανειλημμένα είπε ότι πέρα από αυτά τα 41,8 δις δεν προτίθεται να απορροφήσει άλλα κονδύλια και αν δεν συμβεί κάτι άλλο αυτόματα εκπνέει η συμφωνία στα τέλη του τρέχοντος. και δεν νομίζω ότι θα ζητηθεί περαιτέρω εκταμίευση ή παράταση του προγράμματος ε, μέχρι το τέλος του 13. Αντολίν, ε, θέλεις να επανέλθεις? Όχι, ωραία. Ε, Ευχαριστώ κύριε Ρέγκλινγκ. Έχουμε ξανασυζητήσει το θέμα του ESM και είπαμε ότι θα προτιμούσαμε να είναι κοινοτική η μέθοδος και φαίνονται σήμερα εντυπωσιακά οι συνέπειε. Τα είπε και ο κύριος Γκίγκολτ, σας έκανε τα σωστά ερωτήματα και από τη δική σας αίσθηση και είναι κατανοητό δώσατε ε, τις απαντήσεις σας. Αυτό δεν μπορεί να μας ικανοποιεί. Ε, τι θα συζητήσουμε τώρα για το Ταμείο Εξυγίασης και ε, το ίδιο θέμα θα ξαναμπεί του δημοκρατικού ελέγχου. Ε, εντάξει, ωραία μας τα λέτε, οραματικά και ακούσαμε και τον κύριο Μπαρνιέ για το Ταμείο εξηγήσεις και πού θα πρέπει να ενταχθεί και τα Και ο ίδιος ο κύριος Μπαρνιέ ε, προσωπικά είπε χωρίς να είναι τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά όταν συζητάς κανείς και, έχει ιδέες και οράματα, ε, και μας είπε και μας ότι θα μπορούσε να φανταστεί και την εξυγίαση των τραπεζών, ε, και το Ταμείο το ίδιο να το εντάξουν στον ESM. Δηλαδή προοπτικά στο πολύ απότατο μέλλον θα μπορούσαν να συγχωνευτούν το Ταμείο Εξυγίασης των Τραπεζών μαζί με τον ESM. Αυτό βέβαια χρειάζεται αλλαγή εκβάθρων και τροποποίηση των συνθήκων. Ξέρω ότι σήμερα το πρωί δεν θέλετε και δεν μπορείτε να δεσμευτείτε, το είπατε, που να ε, δεσμεύει ε, πολιτικά ε, τη θέση σας, αλλά από τη σημερινή σας θέση, εσείς με την ιδιότητά σας και με τα καθήκοντα που έχετε, βλέπετε ε, κάπου εμπόδια, δυσκολίες σε ένα τέτοιο δρόμο. Αυτό που είπε ο κύριος Μπαρνιέ εδώ και το σκιαγράφης, έτσι σκεπτόμενος φωναχτά. Γιατί εγώ έχω πολύ μεγάλη συμπάθεια για μια τέτοια πρόταση. Εσείς πώς τη βλέπετε. Δεν ήξερα ότι ο κύριος Μπαρνιέ έχει τέτοιες προσωπικές απόψεις. Ενδιαφέρον μου φαίνεται. Ε, έχω ακούσει και από άλλους ότι κυκλοφορεί αυτή η ιδέα σε κάποιους κύκλους. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχουν συνέργειες για τον ESM. Για ποιο λόγο να αναλάβει αυτό το ρόλο. Αυτός ο ρόλος που έχουμε τώρα έχει να κάνει με χρηματοδότηση και διάφορους τύπους. Ε, χρηματοδότησε ε, λειτουργίες τύπου Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και έχουμε και πολλή δουλειά και η άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι κάπως διαφορετικό αυτό και ως κλάδος και χρειαζόμαστε να προσλάβουμε και ειδικό προσωπικό που θα εποπτεύσει στην αναδιάρθρωση των τραπεζών. Για να πάμε στην εξυγίανση χρειάζεται επίση ε, διαφορετική ειδίκευση. Πού είναι η συνέργεια. Δεν είναι συναφή τα αντικείμενα. Αν με ρωτάτε ε, μακροπρόθεσμα την προσωπική μου άποψη, όπως σας είπα και προηγουμένως, Βλέπω να μπαίνει στη συνθήκη ο ESM να γίνεται ε, θεσμικό όργανο, δεν ξέρω πότε, μακροπρόθεσμα έτσι το φαντάζομαι και εκεί θα χρειαζόμαστε μια διαφορετική δομή, ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο για την εξυγίαση των τραπεζών και μακροπρόθεσμα για την εποπτεία των τραπεζών. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέκαθεν έλεγε ότι δεν ε, ε, δέχεται αυτό το ρόλο με μεγάλο ενθουσιασμό, θα προτιμούσε ένα ξεχωριστό θεσμικό όργανο, αλλά βραχυπρόθεσμα κατανοούν ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, οπότε με βαριά καρδιά το δέχονται, αλλά το ιδεώδες θα ήταν να υπάρχει ένα διαφορετικό θεσμικό όργανο για κάθε μια από τις διαφορετικές αυτέ αυτές λειτουργίες και για την εξηγέση των τραπεζών. Βέβαια, πώς πάμε μέχρι εκεί. Γι' αυτό έχουμε το SSM τώρα που μπαίνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλαμβάνει, αλλά γενικά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας δεν προσφέρεται να αναλαμβάνει τέτοια καθήκοντα. Ε, για να πάμε από εδώ μέχρι εκεί, <laughs> Οι Ιρλανδοί θα λέγανε εγώ δεν θα άρχιζα από εδώ και μάλλον αυτό πρέπει να, πούμε κι εμείς. Λοιπόν υπάρχουν διάφοροι που έχουν κολλήσει σε άλλες επιτροπές. Ε, θα, έχουμε, θα έχουμε χρόνο για τους συναδέλφους, το έχω ήδη υποσχεθεί στην Ελίζα. Για πάμε στο Θεόδωρο τώρα. Thank you very much. Ε, ε, ε. Ευχαριστώ. Ε, συγγνώμη, θα εστιάσω την παρέμβασή μου στην Ελλάδα βλέπουμε την ε, μονάδα εργασία ε, που πέφτει και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Η μεγαλύτερη, από, ε, μία, από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες, η Βιοχάλκο, αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να μεταφέρει την έδρα της από την Ελλάδα στο Βέλγιο. 15% των ελληνικών εξαγωγών έχει αυτή η εταιρεία. Ταυτόχρονα όταν τους ε, ρωτήσαμε μας είπαν ότι το κόστος χρηματοδότησης ε, για μια επιχείρηση στην Ελλάδα είναι κάτι το ανέφικτο, είναι, ε, ξεπερνά πάνω από τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες, αυτό πληρώνουν οι Γερμανοί παραδείγματος χάρη. Και ρωτώ, Α, όχι. Να πω επίσης ότι Πέρα από το πετρέλαιο, ε, το πρώτο εξάμεινο ε, έχουν πέσει οι εξαγωγές μας επίσης λόγω του προβλήματος χρηματοδότησης στον ιδιωτικό τομέα. Το 2012 τώρα ε, είχαμε γενικές κρατικές δαπάνες, το 15% του ΕΑΕΠ που χρηματοδοτούνται εν μέρη ε, ε, από χρήματα άλλων μέσω του ESM και ταυτόχρονα ε, έχει εκμηδενιστεί ο ιδιωτικός τομέας λόγω του, της διαφοράς επιτοκίων και όλα τα υπόλοιπα αλλά η διαφορά στα επιτόκια έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί δεν γίνεται να λειτουργήσει μια επιχείρηση με 10% επιτόκιο σε ευρώ. Ε, πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση στο εγγύς μέλλον. 1,4 εκατομμύρια είναι άνεργοι. 28% του εργατικού δυναμικού. Πώς μπορούν να βρουν απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα όταν εκείνος καλείται να αντιμετωπίσει ένα 10% επιτόκιο. Πώς. Θα προσπαθήσω ε, να είμαι πολύ προσεκτικό στην παρέμβασή μου. Θα κάνω μια διαφοροποίηση ανάμεσα στην πρόοδο σχετικά με τους πρόορους δείκτες ε, που παρακολουθούν ε, εκ του το ψηφιακές αγορές και να το διαφοροποιήσω από αυτό που νιώθουν οι πολίτες. Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση. Έχουμε λοιπόν τους δείκτες, ε, ανταγωνιστικότητες, τρέχοντες λογαριασμοί. Αυτά χρειάζονται, πρέπει να έχουμε τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Πρωτού δούμε τα ωφέλη. Είναι ατυχές, αλλά ε, έτσι συνέβαινε ανέκαθεν Του τελευταίους αιώνες στην οικονομική ιστορία όλων των εθνών υπάρχει καθυστέρηση και τίμημα τίμημα που επομίζεται η Ελλάδα γιατί το εφαλτήριο, η αρχική της θέση ήταν πολύ δυσχερέστερη σε σχέση με αυτή των άλλων χωρών που ε, απευθύνθηκαν στο EFSF και ESM και ως εκ τούτου ε, η προσαρμογή είναι πιο επώδυνη και χρονοβόρα. Ε, όντως, είναι σημαντική η βελτίωση των δικτών, ανταγωνιστικότητα. Ε, οι τιμές αρχίζουν να πέφτουν όχι επαρκώς, πάλι υπάρχει χρονοκαθυστέρηση γιατί η ευελιξία της οικονομίας δεν είναι τόσο καλή. Αν τη συγκρίνουμε με την Ιρλανδία, οπότε ε, για να περάσει αυτή η μείωση του, της μονάδας κόστος εργασίας και να φανεί στις τιμές ε, πρέπει να περάσει καιρός. Ε, η δημοσιονομική προσαρμογή, η κυκλική προσαρμογή, 3% τα τελευταία χρόνια ε, συγγνώμη, 12% σε τρία χρόνια βελτιώνεται η ίσπραξη φόρων, αλλά ε, ε, η δημοσιονομική εξυγίανση όντω είναι δύσκολη γιατί το 2008-2009 ήμασταν στο 15% του ΕΑΕΠ. Έπρεπε οπωσδήποτε να μειωθεί. Οι συνθήκες χρηματοδότησης της χώρας ε, είναι δύσκολες διότι δεν υπάρχει επαρκής εμπιστοσύνη για να επέμβει ο ιδιωτικός τομέας με τη χρηματοδότηση ως μέρος του ε, μνημονίου ε, καταβάλει τώρα η Ελλάδα ε, τις καθυστερούμενες οφειλές. Αυτό δημιουργεί ρευστότητα. Ακολουθούμε τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είναι η πιο δύσκολη υπόθεση. Η Ελλάδα έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι το ζουν καλύτερα. Ε, και χωρίς το EFSF και ESM θα ήταν ακόμη δυσκολότερη η προσαρμογή. Η χρηματοδότηση από το ESM και από το δούνου του σημαίνει ε, ότι μπορεί να μοιραστεί η προσπάθεια σε μια σειρά ετών, αλλιώς θα έπρεπε άμεσα να γίνουν όλα και αυτό θα ήταν σίγουρα χειρότερο. Ευχαριστώ. Ε, περώτηση είναι, αλλά αυτό που πραγματικά ερωτώ είναι για ποιο λόγο υπάρχει ανισορροπία για την προσαρμογή ανάμεσα ε, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα, διότι αυτή τη στιγμή όλοι οι άνεργοι, 99% των ανέργων ε, είναι στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί υπάρχει αυτή η ανισορροπία. Ε, ο ιδιωτικός τομέας θα μας βγάλει από την κρίση, αυτό ελπίζουμε, και όμως εκείνος πλήττεται περισσότερο. Αυτό είναι το πραγματικό μου ερώτημα. Ε, απάντηση. Νομίζω ότι οι περισσότερε μεταρρυθμίσεις προκύπτουν από το μνημόνιο που υποπτεύει η Τρόικα θα οδηγήσουν σε μια κατάσταση όπου θα υπάρξει μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για τον ιδιωτικό τομέα. Συρρυκνώνεται ο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, αυτό είναι προφανέ. και ο ιδιωτικό τομέα με την απορρίθμιση θα έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, να μεγεθυνθεί και να δημιουργήσει θέσει απασχόληση. Ε, σωστά περιγράψατε τα προβλήματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ενθαρρυντικό που ο ΣΑ στην ετήσια έκθεση που κάνει για τι μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη του ΩΣΑ. Ξέρετε ότι πάμε από την Κορέα μέχρι το Μεξικό και είναι εκεί όλες οι βιομηχανοποιημένες χώρες. Η Ελλάδα είναι πάνω-πάνω στον κατάλογο σε σχέση με τον αριθμό των μεταρρυθμίσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή, σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα του ΩΣΑ. Ε, αυτό μας λέει ότι θα έπεται και άλλη πρόοδος, αλλά προς το παρόν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική εξυγίανση βαρύνουν τους ώμους του πληθυσμού στην Ελλάδα και τα πράγματα ήταν χειρότερα πριν από τέσσερα χρόνια. Είναι χρονοβόρα και ιδιαίτερα επώδυνη, ξαναλέω, προσαρμογή, αλλά σας είπα τι λέει ο ΣΑ, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στην πράξη. Ε, ε, ε λυπάμαι που ε, έφυγε ο κύριος Κλίντς γιατί το συζητήσαμε μακρόν το ζήτημα στο Βίλνιους. Ε, συμβαίνουν πάντως ε, αυτά που επιθυμούμε, είναι αργή η πρόοδος, αλλά το μόνο που έχουν να κάνουν οι άνθρωποι να περιμένουν τα καλά αποτελέσματα. Ελίσσα, σου ξαναδίνω το λόγο, ζητώ συγγνώμη που περίμενες τόση ώρα. Ναι, θα μιλήσω αγγλικά. Θέλω να επανέλθω στο ζήτημα των προαπαιτούμενων που ζητάει το ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των τροπεζών. Αντιλαμβάνουμε ότι πρώτα γίνεται bail-in και αν χρειαστεί μετά θα είστε έτοιμοι να ανακεφαλαιοποιήσετε μια τραπεζά. Όμως, το εκείνο τη στιγμή το Ταμείο Αναχρηματοδότησης θα έπρεπε να, ε, θα έπρεπε να επέμβει. Και όπως είπε και ο συνάδελφος, αν μας λέτε ότι δεν μπορούμε να ενισχύσουμε το ταμείο, γιατί αυτό χρειάζεται μεταρρύθμιση της ε, συνθήκης, τότε πώς και πού το ESM εντάσσεται και επεμβαίνει στην διαδικασία εξηγήσης. Με αυτό είναι τι, σε τι σχέση με το Ταμείο Εξυγίανσης. Θα υπάρχει ανταγωνιστική σχέση, θα υπάρχει συμπληρωματική σχέση και χρονικά αυτό πώς θα γίνεται, πότε. Πριν ή μετά την επέμβαση του Ταμείου Εξυγίανσης. Σε πρώτο ερώτημα και δεύτερο. Εάν δημιουργηθεί αυτός ο ενιαίος μηχανισμός εποπτείας. Εγώ είχα αντιληφθεί ότι αυτό θα επέτρεπε στο ESM να επεμβαίνει χωρίς να υπάρχει εγγύηση από την κυβέρνηση του κράτους μέλους στον οποίο εδρεύει το πιστοτικό ίδρυμα. Γιατί πλέον θα έχουμε έναν ενιαίο μηχανισμό. Άρα υποτίθεται ότι θα υπάρχει εμπιστοσύνη προς αυτόν. Αλλά από την απάντηση που μου δώσατε κατάλαβα ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να συνεχίσουν να εμπλέκονται ως ε, εγγυητές του δανείου. Μήπως θα μπορούσατε να μου το διευκρινίσετε αυτό. Ναι, για το πρώτο σας ερώτημα. Δεν έχουν διευκρινιστεί όλες οι λεπτομέρειες. Γι' αυτό οι Υπουργοί Οικονομικών του Eurogroup της Ευρωζώνης αποφάσισαν να μην καθορίσουν, να μην οριστικοποιήσουν τις ε, προβλέψεις ε, για την εξυγίαση των τραπεζών, των BRRD, μέχρι να, να συμφωνηθεί το BRRD. Άρα αυτά τα δύο θα πρέπει να γίνουν μαζί. Δεύτερον, όσον αφορά την επέμβαση των κρατών μελών για εξυγένση, σε εκείνη την περίπτωση το ESM δεν θα επενδύει σε ε, αφαιρέγγιες τράπεζες, το οποίο σημαίνει ότι ο λόγος ε, ε, κεφαλαίων θα είναι 4 προς 1 προκειμένου να... Και το ESM θα παρεμβαίνει προκειμένου να αυξήσει αυτόν τον λόγο κεφαλαίων προς το 4 προς 1 ή 9 προς 1 ό,τι χρειάζεται. Πάντως οι λεπτομέρειες θα πρέπει να διευκρινιστούν στο μέλλον και σε καμία περίπτωση δεν θα θέλαμε μια ανταγωνιστική σχέση με το ταμείο. Αυτό δεν, θα, ε, δεν συμφέρει κανέναν ευελπιστώ ότι αυτά τα ερωτήματα θα διευκρινιστούν τους επόμενους μήνες. Για τη δεύτερη ε, ερώτησή σας για το μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης, ε, αυτή τη στιγμή σε αυτό εγκριθεί δεν θα υπάρχει πλέον εγγύηση από την πλευρά των ε, κρατών. Ε, αυτή τη στιγμή θα αξιοποιείται λοιπόν αυτό το μέσο άμεσης ανακεφαλαιοποίησης για μια, ένα πιστοτικό ίδρυμα. Δεν θα χρειάζεται πλέον η εγγύηση του κράτους στο οποίο εδρεύει. Εξάλλου, αυτό το ήταν στην βάση του προβληματισμού που μας οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρέπει να διακόψουμε, να σπάσουμε αυτή τη σχέση μεταξύ των, ε, των χρεών των τραπεζών και του κρατικών χρεών τελικά. Ευχαριστώ. Έχω και άλλη ερώτηση για την κατάσταση στις χώρες υποπίεση, χώρες όχι τράπεζες. Εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας. Είμαι λιγότερο αισιόδοξη, αν και χάρηκα που άκουσα να είστε εσείς τόσο αισιόδοξο. Τι να υποθέσω αυτά που είπατε, ότι ε, στην Πορτογαλία δεν θα χρειαστεί και άλλο πακέτο διάσωσης και ότι η Πορτογαλία δηλαδή μπορεί να ακολουθήσει την ίδια τραπό με την Ιρλανδία και να διαπραγματευτεί ε, κάποια πιστοτική γραμμή μεταβατική για να βγει από αυτή την κατάσταση. Και δεύτερη υποσημείωση, η σχέση μεταξύ των δικών σας απαιτήσεων για το Ταμείο και ο τρόπος συνεργασίας με την Τρόικα. Εσείς συζητάτε με την Τρόικα ποτέ αν οι συστάσεις μπορούν να βελτιωθούν γιατί δεν έχουν δουλέψει όταν είναι διαφορετικά τα αποτελέσματα από αυτά που ε, προέβλεπαν. Εσείς πώς συνεργάζεστε με την Τρόικα σε αυτά τα προγράμματα και στη χρηματοδότησή σας. Ελπίζω αυτό που ονομάζεται αισιοδοξία να είναι ρεαλισμός από πλευράς μου. Μακάρι. Ε, και, δηλαδή να δικαιωθώ. Και στην Πορτογαλία οι πρώιμοι δείκτες μας δείχνουν ότι έχει γίνει καλή πρόοδος. Δεν είναι το τέλος του δρόμου, ούτε η κρίση πέρασε. Ο κόσμος δεν βλέπει την πρόοδο, αλλά ε, γνωρίζετε στις ε, τρέχουσες συναλλαγές είχε τεράστιο έλλειμμα η Πορτογαλία ε, και έχει εξαφανιστεί. Για πρώτη φορά έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Το ξέρω ότι ο λαός δεν το νιώθει αυτό ακόμα. Τι θα γίνει του χρόνου όταν ε, τελειώσει το τρέχον πρόγραμμα. Είναι πολύ νωρίς ε, για μένα να πω τι θα συμβεί. Θα εξαρτηθεί από τις εσωτερικές εξέλιξεις στην Πορτογαλία, αλλά και από τις εξωτερικές. Εάν πετύχουν οι γειτονικέ χώρες και αν ανθεί το παγκόσμιο εμπόριο, θα είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από ότι αν υπάρχουν προβλήματα γενικότερα στην παγκόσμια οικονομία είναι αλληλένδετα. Αυτό εν μέρη το ελέγχει η πορτογαλική κυβέρνηση και εγώ δεν μπορώ παρά να τους ενθαρρύνω να συνεχίσουν στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που δεν ελέγχουμε και θα είναι αποφασιστικά. Ε, ε, οποιοςδήποτε ισχυρίζεται ότι μπορεί από τώρα να προβλέψει θα χρειαστεί, δεν είναι σοβαρός στι προβλέψει. Χρειάζεται να περιμένουμε λίγο παραπάνω. Η σχέση μας με την Τρόικα. Γνωρίζετε ότι η Τρόικα είναι αρμόδια ε, για τις διαπραγματεύσεις με τις χώρες ως προς τα προαπαιτούμενα. Για τα συγκεκριμένα μέτρα δηλαδή που έχουν επιπτώσεις και στους λαούς και στις χώρες. Εμείς δεν αποφασίζουμε. Συμμετέχουμε μεν γιατί τελικά θα πρέπει να εξηγήσουμε αν μπορούμε να δώσουμε τη χρηματοδότηση ή όχι και ποια θα είναι τα στάδια και συνοδεύουμε τη διαδικασία αυτή για να ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Αλλά εμεί δεν αποφασίζουμε για την προσαρμογή ούτε ποιε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι πιο σημαντικές ή πιο επίγουσες. Μπορεί να έχουμε τη γνώμη μας καμιά φορά, ιδιαίτερα στα τραπεζικά συμμετέχουμε γιατί έχουμε και κάποια πραγματογνωμοσύνη εκεί, αλλά για τα προαπαιτούμενα και τους όρους αυτά είναι θέματα της Τρόικας και δική της ευθύνη. Ωραία. Ε, ε, εγώ, ο Σβέν και η Άννη αρκούμε για να συμπληρώσουμε το χρόνο που μας μένει. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Είπατε στην εισαγωγή σας ότι η Ιρλανδία, για παράδειγμα, ε, βγαίνει στην αγορά κρατικών ομολόγων με λογικό επιτόκιο, 4%. Αυτό τι σημαίνει. Είναι πιο φτηνό από αυτό που πληρώνει για τα δάνεια η FSF. Ποια είναι η σχέση τώρα, ε, ποια είναι ε, τα επιτόκια που πληρώνει στο δάνειο του UFSF σε σχέση με τα κρατικά ομόλογα. Υπάρχει κάποιο τιμωρητικό στοιχείο εδώ. Δεν το έχω καταλάβει. Βασικά πληρώνουν το κόστος και δεν υπάρχει πλέον αυτό το, το τιμωρητικό. Όταν δημιουργήθηκε ο EFSF πριν από τρία χρόνια, αρχικά υπήρχε ένα τέλος ε, επιπρόσθετο, μια προσάυξηση για να αποτραπούν ε, οι ενδιαφερόμενοι. Όμως ε, το κύριο Κρουπ συνειδητοποίησε ότι η βιωσιμότητα είναι το ζητούμενο και μείωσε το κόστος ούτως ώστε να επιτύχουμε βιωσιμότητα. Οπότε στους οφειλέτες μας ε, ε, χρεώνουμε ακριβώς ε, αυτό που πληρώνουμε εμείς με κάποιες μονάδες βάσης επιπρόσθετες για τα λειτουργικά τα, από τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα παίρνουμε από τις αγορές ορισμένες φορές για τα εξάμεινα, παραδείγματος χάρη έχουμε αρνητικά επιτόκια και οι χώρες προγράμματος ε, εποφελούνται από αυτό. Οπότε αυτό που κάνουμε είναι ότι κάθε μέρα υπολογίζουμε ένα μέσο επιτόκιο, δηλαδή ε, ε, ο μέσος όρος είναι 2 με 2,5%. Ορισμένες φορές αυξάνεται. Τα βάζουμε όλα πάντως σε ένα κοινό κορβανά. Ε, αν δείτε τα δεκαετή κρατικά ομόλογα, βλέπετε πόσο υποφελώς είναι αυτό για την Ιρλανδία. Και το βραχυπρόθεσμο είναι βέβαια, γιατί είναι 4%, αλλά είναι ευνοϊκή η όρη για την Ιρλανδία. Ακόμη ευνοϊκότερη εννοείται για την Ελλάδα και για την Ιρλανδία, διότι ε, βρίσκονται ε, με υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης. το δούνο του είναι 3%, είναι πολύ φθηνότερο, αλλά εμεί έχουμε μεγαλύτερη περίοδο ρήμανση, οπότε είναι σημαντικά τα ωφέλη ε, για αυτές τις χώρες. Ε, εγώ, λέει η Πρόεδρος, θυμάμαι ότι άσκησε πίεση εδώ το Κοινοβούλιο, ειδικά η Επιτροπή μας, ε, για να, έχουμε αυτό, να αρθεί αυτό το τιμωρητικό στοιχείο αρκετά νωρί στη διαδικασία Σβέν. Ευχαριστώ πολύ Να Έχω και άλλη ερώτηση κύριε Ρέγκλινγκ ως προς την έννοια της βιωσιμότητας του χρέους για την Ελλάδα αλλά και για τα άλλα προγράμματα μπορεί κανείς να προβληματίζεται για το πώς στην πράξη λειτουργεί αυτό. Στο ΚΙΕΛΟ υπάρχει το Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Οικονομία με ένα βαρόμετρο για το χρέος υπολογίζει ότι η Ελλάδα αν επανέλθει στο 2% ανάπτυξης χρειάζεται 14% ε, πλεόνασμα. Εάν είναι 4% η ανάπτυξη που είναι ανεδαφικό αυτό γιατί θα χρειαστεί μεγάλο χρόνο χρειάζεται πάνω από 10% πλεόνασμα. Αλλά πάνω από 5% πλεόνασμα του ΑΕΠ δεν υπάρχει πουθενά εδώ και καιρό. Πόσο μάλλον στις δυτικές ε, βιομηχανικές χώρες. Με άλλα λόγια, αυτό το θέμα της βιωσιμότητας του χρέους δεν παραβιάζεται και μάλιστα κατάφορα και στους κανόνες σας έχετε και εσείς αυτό και τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλουμε πρώτον για την αξιολόγηση ε, των δανείων που δίνονται ε, και επίσης τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς για το πώς μεταφέρεται στην πράξη η βιωσιμότητα του χρέους και λειτουργικά πώς ε, δουλεύει. Ε, δηλαδή ε, παρατείνεται, ε, τραβάει σε μάκρος μια διαδικασία πτώσευσης. Στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν και άλλες οικονομίες, συζητιέται ένα κούρεμα, αλλά μπορεί να υπάρξει και μια τρίτη εκδοχή που είναι η φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας και η μεγάλη ιδιωτική περιουσία που δημιουργήθηκε σε καιρούς παχιών αγελάδων μπορεί να αξιοποιηθεί. Ε, εσείς πώς το βλέπετε αυτό για τις μεταρρυθμίσεις της χώρας κρίσης. The um, and how to manage and how to achieve that's... Το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους είναι σίγουρα σημαντικό. Τώρα φιλοσοφικά και από πλευρά οικονομολογική είναι δύσκολο γιατί υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Μας δώσετε ένα παράδειγμα με ρυθμό αύξησης 2%-4% και πόσο μεγάλη διαφορά ε, προκαλεί αυτό. Δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να προβλέψουμε ακριβώς ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης σε αυτές τις χώρες. Ε, πολλές φορές δυσκολευόμαστε ακόμα και την επόμενη χρονιά να προβλέψουμε ποιος θα είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Επομένω, ε, είναι ανεδαφικό να πιστεύουμε ότι μπορούμε να προβλέψουμε την ανάπτυξη ε, κατά τη διάρκεια δέκα ετών. Εγώ θα ζητούσα να μην μιλάμε για μια παρατεταμένη χρεοκοπία, γιατί αυτή είναι μια ορολογία την οποία χρησιμοποιούν ε, κάποια άλλα μέλη ε, δεν λέω ότι είναι νομοτέλεια, αλλά περιγράφω. Ε, προσοχή, στην περιγραφή να είμαστε σαφείς περί τίνος πρόκειται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά όταν ισχύει κάτι το περιγράφουμε. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Είναι δύσκολο, αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να έχει βεβαιότητες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, όλα και εμείς, ε, κάνουμε σενάριο, ε, σενάρια και μελετούμε τη βιωσιμότητα. Ένα πολύ βασικό σημείο που συχνά παραμελείται και από το Ινστιτούτο για την Παγκόσμια Οικονομία του Κιέλου είναι ότι τεράστια διαφορά αν έχεις 100 ή 120% του ΑΕΠ ε, ως χρέος που είναι συνήθως ο στόχος να υπερβαίνει το 120% το χρέος σε ορίζοντα δεκαετίας είναι διαφορετικό από το επιτόκιο ε, το οποίο χρηματοδοτείται. Μιλήσαμε για το δικό μας επιτόκιο και είναι τεράστια διαφορά εάν μια χώρα σαν την Ελλάδα θα πρέπει να χρηματοδοτεί το επίπεδο χρέους της σε επιτόκια αγοράς που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι 8% μέχρι 6% ενδεχομένω να μειωθεί ή αν χρηματοδοτείται με 1,5-2% που μας πληρώνουν εμά. Και εμείς ε, χρηματοδοτούμε για 30 χρόνια. Είναι τεράστια διαφορά αυτή. Μπορεί κανείς να έχει πιο ψηλό επιτόκιο αλλά όταν είναι χαμηλό το επιτόκιο μπορεί να είναι πιο μακροχρόνιο το δάνειο, αυτό που δείχνει η Ιαπωνία. Δηλαδή ε, εφαρμόζουμε στην Ελλάδα οι ιαπωνικές συνθήκες για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα που είναι ε, πολύ μεγαλύτερο από ε, οποιαδήποτε άλλα παραδείγματα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να είναι βιώσιμο. Κανείς δεν έχει, δεν διεκδικεί εδώ το αλάθητο. Ούτε μπορούμε να πούμε αν η Ελλάδα πρέπει να φτάσει στο 120% το 2020, το 2022 και οτιδήποτε παραπάνω ε, είναι καταστροφή, οτιδήποτε πιο κάτω σημαίνει έξοδο στις αγορές. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι, δεν υπάρχει καμία μέθοδος που να το υπολογίζει με ακρίβεια, αλλά αν δούμε τις συνθήκες, αυτό που βοηθάει τις χώρες που δανείζονται από τον ESM και το FSF είναι ότι μεγάλη οριμότητα, χαμηλά τα επιτόκια και αυτό μας δείχνει και μας δίνει τη βεβαιότητα ότι με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις κανονικά θα πρέπει να είναι σε θέση σε αυτό το χρονικό διάστημα να φτάσουν σε βιωσιμότητα. Ευχαριστώ. Γιάννη Ποδηματά, παρακαλώ. Επιτρέψτε μου να παρέλθω σε κάποια πιο επίγουσα σημασία θέματα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι η Ελλάδα ε, εκτιμά τις δανειοδοτικές ε, συνθήκες ε, που προσφέρει το ESM στην Ελλάδα, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Κυλακάκης και εσείς είπατε επίσης ότι η σημαντικότερη πρόκληση για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι να ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της και πράγματι έχετε δίκιο. Κάτι... Οι μεταρρυθμίσεις, οι δομικές μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο και γι' αυτό τα αποτελέσματα του προγράμματο δεν μπορούν να είναι ακόμα ορατά από τους πολίτε. Ε, σωστά επίσης είπατε ότι το σημείο εκκίνησης της Ελλάδας ήταν ε, πιο δυσχερές από άλλες χώρες. Όμως το ζήτημα είναι τελικά πότε θα μπορέσουμε να δούμε μια βελτίωση την οποία θα τη δουν οι ίδιοι οι πολίτες. Ε, το, το, το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα με μένα περισσότερο είναι πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι δεν θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση της κατάστασης. Η έλλειψη χρηματοδότησης στον ιδιωτικό τομέα οδηγεί τις ελάχιστες εναπομείνουσες ιδιωτικές επιχειρήσεις να εγκαταλείψουν τη χώρα και να ε, μεταφέρουν την έδρα τους στο εξωτερικό γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν χρηματοδότηση ή ε, εν πάση περιπτώσει χρηματοδότηση με λογικά επιτόκια εντός της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν κίνδυνο περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομικής ε, κατάστασης της χώρας. Γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος ο κ. Σκυλακάκος Χάλκο, ε, το 15% καλύπτει το 15% των εξαγωγών. Για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά μας πρέπει να ενισχύσουμε τις εξαγωγές, αλλά οι εξαγωγικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν τη χρηματοδότηση που χρειάζονται. Και μπαίνουμε έτσι σε ένα φαύλο κύκλο που θα οδηγήσει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από την ήδη δύσκολη που ε, βιώνουμε. Είναι πραγματικό το πρόβλημα που περιγράφεται. Είναι, υπάρχουν δύο σημαντικά στοιχεία στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας που συμφωνηθήκε με την Τρόικα και προσπαθεί να ρυθμίσει αυτά τα προβλήματα. Πρώτον, αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών και ε, ε, διαρκή είμαστε στο μέσο της διαδικασίας σε σχέση με την εκταμείευση του FSF προς την κυβέρνηση. 15 δις από αυτό το ποσό έχουν εκταμιευθεί, έχουν ε, ήδη ε, διοχετευτεί για την Ελλάδα. Αυτό εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα και ε, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στο HFSF. Ε, και χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων μεγαλύτερων ε, τραπεζών ούτω ώστε να παίξουν το ρόλο που πρέπει στην πραγματική οικονομία ως χρηματοπιστωτικοί διαμεσολαβητές ενδιάμεση ε, επιστρέφοντας έτσι σε πιο φυσιολογικές οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα. Ένα άλλο σημαντικό σημείο και ακροφυγώς το ανέφερα, ως μέρος αυτού του προγράμματος μεταρρυθμίσεων το ελληνικό ε, κράτος ε, τώρα καταβάλει ε, τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, απεφεύγοντας την πραγματική αποτελμάτωση της οικονομίας, διότι έχουν προσφέρει υπηρεσίες σε κάποιοι, αλλά πρέπει να αποζημιωθούν, δεν μπορούν να αποπληρώσουν συνέχεια τις τράπεζες, είναι ένας φαύλος κύκλος και δυσκολεύει τα πάντα. Ε, έχει αρχίσει να πληρώνει λοιπόν ε, αρκετά δισεκατομμύρια ήδη η ελληνική κυβέρνηση σε καθυστερούμενες οφειλές. Αυτό θα βοηθήσει την οικονομία. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές, αλλά δεν αυξάνονται τουλάχιστον, μειώνονται πλέον. Εάν συνεχιστεί αυτό και έχουν αποπληρωθεί όλα, τότε σε μεγάλο βαθμό θα ανακουφιστούν οι, οι επιχειρήσεις που έχουν αξιώσει ενώπιον του δημοσίου, διότι έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους και επιστρέφουμε έτσι στην ομαλή κατάσταση όπου θα χορηγούνται δάνεια και άρα θα υπάρξει μια ανακούφιση χάρη σε αυτές τις κοινές ελληνικής κυβέρνησης. Ε, πρόεδρος, ωραία, σας ευχαριστούμε. Πολύ χρήσιμα όλα αυτά. Ε, και ελπίζουμε να είναι πλέον τακτικές οι επισκέψεις σας και να μπορέσουμε να έχουμε ένα ε, τέτοιο χρονοδιάγραμμα συνεργασίας ε, και να συνεχίσει ο ESM να διαδραματίζει αυτό το τόσο σημαντικό ρόλο για την σταθερότητα της Ευρωζώνης και της επερχόμενης Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ένωσης. Ευχαριστούμε. Τα λέμε το απόγευμα.